Mes chers collègues, je vous propose μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Θα είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Με βεβαρημένη μερίσια διάταξη. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, παρακαλώ λίγη ησυχία καταρχάς. Θα ήθελα να αποτέσω φορά τιμή σε έναν συνάδελφό μα. ο οποίος δυστυχώ απεβίωσε. Η οικογένειά του, η Επιτροπή Προπολογισμών, πραγματικά έχει θλιβεί βαθύτατα, διότι χάσαμε το φίλο μας Πόρτας καταρχάς. Πριν από δύο ημέρες ο κύριος Γύρι Χάβελ επίσης απεβίωσε, όπως μάθαμε πριν από δύο ημέρες. Ήταν 54 ετών, Τσέχος, μέλος της σοσιαλιστικής ομάδας και πρόεδρος της Τσέχης Αντιπροσωπείας στην ομάδα. Αντιπρόεδρος δε της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις της Ένωσης με την πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ήταν μέλος και της Επιτροπής μας αλλά και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Δυστυχώς όμως ε, είχε μια βαρύτατη ασθένεια τα τελευταία χρόνια έτσι και δεν μπορούσε συχνά να συμμετέχει στις συνεδριάσεις μας. Προτείνω στον ε, Γκέραν Φέρμο να μας μιλήσει για τον ε, Γεριχάβελ και μετά θα τηρήσουμε ως λεπτούς υγιή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πριν από λίγε μέρε πράγματι λάβαμε τα πολύ δυσάρεστα νέα τα απεβίωσε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω τη ασθένειά του δεν ε, μπορούσε να ε, πεί σε αεροπλάνο, δεν μπορούσε να έρθει εδώ στι Βρυξέλλε. Στο Στρασβούργο όμω πάντοτε ήταν παρόν και την τελευταία φορά που τον συνάντησα στο Στρασβούργο ήταν ιδιαίτερα ε, βαριά, αλλά περιμέναμε ίσω κάτι να, θετική, ε, να θετικά, δεν έγινε. Ήταν οικονομολόγο, πρώην Υπουργό Οικονομικών στη Τσεχική Δημοκρατία, διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στη Τσεχική Δημοκρατία κατά τη μεταβατική περίοδο μετά τον κομμουνισμό και είχε τη φιλοδοξία να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ όμω λόγω τη ασθένειά του δεν κατέστη αυτό ποτέ δυνατό. Δεν μπόρεσε να αναπτύσσει το ρόλο που ήθελε. Στη δική μα ομάδα εσωτερικά ήταν πολύ σημαντικό επίση γιατί είχε ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις, ε, ήταν ε, ιδιαίτερα ε, προσυλλομένος στα θέματα της οικονομικής κρίσης, των οικονομικών κανονισμών και ούτω καθεξής και πραγματικά είχε μεγάλες φιλοδοξίες και πολύ υψηλές γνώσεις για τα οικονομικά ζητήματα. Θα μας λείψει σε όλους και βέβαια η συμπάθειά μας και τη συλληπιτήριά μας είναι στην οικογένειά του. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Γκέρ. Φυσικά όλοι εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, ε, την ε, ε, θλίψη μας προς την οικογένεια και τους φίλους του Γύρι Χάβελ. Παρακαλώ να τηρήσουμε τώρα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κυρίου Γύρι Χάβελ. Σε Σα ευχαριστώ. Ε, σε έχει mm. Έχω και μια άλλη ανακοίνωση, λιγότερο δυσάρεστη. Από σήμερα και μετά ε, θα έχουμε ένα νέο μέλο ε, στην Επιτροπή μα, τον κύριο Νίλ Στόρβαλτ, ο οποίο αντικαθιστά τον πρώην συναδελφό μα, τον Καρ Χάγκλουντ, ο οποίο έγινε υπουργό άμυνα στη Φιλανδία. Ο κύριο Στόρβαλτ είναι εδώ, Καλώς ορίσατε κύριε συνάδελφε. Έχω ήδη συναντήσει τον ε, συνάδελφο Κάρλ Χάγκλουντ τώρα, ήταν συντονιστής ε, των φιλελευθέρων και χάρη στη, στα προσόντα του σε μια, χώρα που στη, σε μια ηλικία που στη χώρα μου άντε και να έχουμε αποκτήσει δικαίωμα ψήφου έγινε υπουργό Άμυνα και πραγματικά του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Επίσης ο αντιπρόεδρος George Lyon ένιωσε μια διαθεσία, ε, υπήρξε ένα ε, μικρό πρόβλημα καρδιακό που αντιμετώπισε, δεν είναι σοβαρό, αλλά ε, νοσηλεύεται και δεν μπορεί να έρθει στη συνεδρίασή μας. Φυσικά φαντάζομαι θα ευχηθώ εκ μέρους όλων μας γρήγορη και καλή ανάρρωση στον George Lyon. Α, στο γιο Λάινεν θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά σημείο ένα της μέσης διάταξης, η έγκριση μέσης διάταξης, αν θεωρείτε ε, ότι δεν υπάρχουν σημεία, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Θα χρειαστεί να αναβάλουμε κάποια θέματα. Θα σας τα πω με τη σειρά όταν είναι. Έχετε τις ανακοινώσεις τα κόμπου News. Οι εργασίες μας, όπως ξέρετε, πάντοτε μεταδίδονται στο webstream, οπότε αυτό ισχύει και για σήμερα. Σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών συνεδρίαση τη 10 η Μαΐου. Επειδή δεν ήταν εγκαιρω διαθέσιμα τα πρακτικά, αναβάλλεται η έγκριση. Ωστόσο, τα πρακτικά τη συνεδρίασης τη 31 η Μαΐου είναι διαθέσιμα και ο ήθιστε, αν μέχρι τη σημερινή μα συνεδρία δεν υπάρξουν αντιρρήσει, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Σήμερα, τώρα, το μεσημέρι στις 3 έχουμε την ετήσια συνάντηση με την ε, Τρόικα και τους που εκπροσωπούν τους εκτελεστικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα κάποια μέλη της Τρόικας, καθώς και εκπροσώπους άλλων οργανισμών στην αίθουσα. Φαίνεται ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί μας για τον προπολογισμό. Λοιπόν, θα έχουμε βέβαια την ανταλλαγή απόψεων σήμερα το μεσημέρι για το θέμα αυτό, για τους πακεντρωμένους οργανισμούς. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 6 και μετά θα μιλήσω λίγο για το σημείο 5, το σχέδιο υπερπολογισμού 2013 και τα αποτελέσματα του τρομερούς διαλόγου που διεξήχθη στις 9 Ιουλίου. 1 Ιουλίου λοιπόν έγινε ο τρομερής διάλογος και συγκεκριμένα μετά την εξέταση και την ενδεικτική ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην Επιτροπή Προπολογισμού του Σύμβουλου Κόμπουτ και πριν την ψηφοφορία σε επίπεδο Κορεπέρ για το σχέδιο προπολογισμού 2013 εχθές το πρωί. Σε συνθήκες που μου φαίνονται ιδιαίτερως ε, περιεργέ. Δεν θέλω όμως να δώσω τη δική μου προσωπική εντύπωση. Πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές μας ε, για να μας πούν οι ίδιοι πώς εκτίμησαν τα αποτελέσματα. Τζοβάνι Τελαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο τριμερής διάλογος αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε με μια στυλίτευση από μέρους μας των καθυστερήσεων που είχαν χαρακτηρίσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου και που δεν είχαν επιτρέψει στο Συμβούλιο να είναι παρόν με μια πραγματική πολιτική εντολή. Εμείς δώσαμε σαφή εντολή για τον τριμερή διάλογο που δώσαμε και μέσω της Επιτροπής Προϋπολογισμού αλλά και στην Ολομέλεια με 540 ψήφους υπέρ δώσαμε αυτή την πραγματική εντολή. Επίσης, από την άλλη, κάποιοι κάνανε μια εντελώς τεχνική ανάγνωση του κειμένου, αλλά δεν υπήρχε καμία πολιτική απόφαση ούτε στο Κορεπέρ ούτε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αυτά για το Συμβούλιο. Άρα η εκπροσώπηση του Συμβουλίου στο τριμερή διάλογο δεν είχε εντολή ουσιαστικά. Τώρα, στον τριμερή διάλογο. Εντοπίσαμε τις προτεραιότητες, όπως προέκυπταν από την εντολή. Τις αναφέραμε, επιμείναμε. Επίσης τονίσαμε ότι το, η συμπεριφορά του Συμβουλίου δεν ευθυγραμμιζόταν με τα συμπεράσματα της ε, του περσινού έτους. Είχαμε αποφασίσει, όπως θυμάστε από κοινού, να παρακολουθήσουμε τις πληρωμές, κάτι που στην πραγματικότητα δεν συνέβη. Γιατί στη συνάντηση για τις πληρωμές ήταν αποκλειστικά παρούσα η Κομισιόν, ενώ το Συμβούλιο επί Δανέζικης Προεδρίας δεν πήρε μέρος. Δεν θέλαμε τα δεδομένα εκκίνησης για τη συνδιαλλαγή τη φετινή για τον προπολογισμό του 2013 να είναι διαφορετικά μεταξύ των δύο αρχών του προπολογισμού, δηλαδή μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου η ερμηνεία, η ανάγνωση που έκανε το Συμβούλιο και που επιβεβαιώθηκε χθε από την ψηφοφορία στο Κορεπέρ. Είναι μια ανάγνωση, είναι μια ερμηνεία που μπλοκάρει το επίπεδο πληρωμών στο, την αύξηση καλύτερα των πληρωμών σε σχέση με το προϋπολογισμό του 12 στο 2,79% και αυξάνει σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό τις ε, δεσμεύσεις στο 1,27%. Αυτή η ερμηνεία σε σχέση με τις προτεραιότητες που είχαν δοθεί στην εντολή για τον τριμερή διάλογο από το Κοινοβούλιο μου φαίνεται ανεπαρκής για να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε τις ευρωπαϊκές ε, προτεραιότητες και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές στα πλαίσια του διαλόγου και εγώ με τις παρεμβάσεις μου, αλλά και ο πρόεδρος Λαμασούρ με τις παρεμβάσεις του, τόνισαν την ασυνέπεια που υπάρχει, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης και 29 η Ιουνίου και από την άλλη στην ερμηνεία που είχε γίνει από την Κόμπουτ στο προπολογισμό. Όπως είδαμε στο Συμβούλιο στις 28 και 29 του μηνός Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συμβουλίου λέγοντας ότι για να βγούμε από την κρίση χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Και αυτό για, για μας σημαίνει ότι θα πρέπει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να είναι στεναρός για την ανάπτυξη Νόμιζα λοιπόν θα υπάρχουν νέοι πόροι ή ουσιαστικοί πόροι για την ανάπτυξη. Όμως, από την άλλη, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Κόμπουτ και χθε από το Κορεπέρ είναι τελείω διαφορετικά. Κινούνται προς άλλη κατεύθυνση. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη δέσμευση ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει αυτό στις ε, πιστώσεις ε, πληρωμών, δεν υπάρχει στις πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων, δεν υπάρχει γενικά. Επομένως, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ερμηνείες, τις διαφορετικές ερμηνείες που κάνουμε. Από την άλλη, η ερμηνεία που κάνει η Κόμπουτ έρχεται σε αντίθεση και με τη φιλοσοφία του Συμβουλίου, μπορώ να πω. Γιατί οι μεγαλύτερε περικοπές που προτείνονται αφήνουν, αφορούν τον τίτλο 1α. Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, το, την 1β, πολιτικές συνοχής εν μέρη τη 2 και ουσιαστικά την 4, σε μεγάλο βαθμό την 4, δηλαδή τις πολιτικές γειτονίας. Σε σχέση λοιπόν με αυτές τις ερμηνείες, με αυτή την ερμηνεία του Συμβουλίου, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο κατελήφθη εξαπίνης. Εσείς θα θυμάστε τις κατευθυντήρες γραμμές μας, θα θυμάστε τις ε, προτεραιότητές μας, αλλά μην ξεχνάτε και τις κατευθυντήρες γραμμές του Συμβουλίου που μιλούσαν ότι η ανάπτυξη ήταν προτεραιότητα του προπολογισμού του 2013, από την άλλη όμως έχουμε περικοπές. Ακριβώς σε εκείνες τις, ε, τους τίτλους όπου ε, υπάρχουν προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την ανάπτυξη. Σε σχέση λοιπόν με αυτό, στο ανακοινωθέν τύπου που κάναμε με τον πρόεδρο Λαμασούρ, τονίσαμε αυτές τις ασυνέπειες, αυτό το πρόβλημα και είπαμε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες από αυτές που προκύπτουν από την ερμηνεία του Συμβουλίου. Στη δουλειά που θα κάναμε, θα κάνουμε τους επόμενους μήνες και για να κάνουμε αυτή τη δουλειά τους επόμενους μήνες χρειαζόμαστε πολλές διευκρινήσεις. Χρειαζόμαστε νέα στοιχεία. Γιατί αν οι προτεραιότητες που έχουν εκφραστεί στο υψηλότατο επίπεδο του Συμβουλίου είναι η ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχε αποφάσει και στον προπολογισμό από το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν τι βλέπουμε αυτές τι αποφάσεις. Χθε το Κορεπέρ ενέκρινε την απόφαση, την πρόταση της Κομισιόν προϋπολογισμού με τρεις ψήφους κατά από τρεις χώρες που είναι πληρωτές, δηλαδή υπάρχει η αντίθετη ψήφος του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. Μία αποχή της Αυστρίας και θα δούμε ότι... Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με, τις, με κάποιες δηλώσεις που είχαμε ακούσει εσωτερικές, αν θα εκφραστούν και πιο έξω. Πάντως, αυτές οι διαφωνίες δείχνουν ότι υπάρχει μια σχιζοφρενία στο, στο Συμβούλιο. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει η Κόμπουτ στο Συμβούλιο σε σχέση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι έχουν κινηθεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλα η Κόμπουτ και άλλα λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ε, μέρες τι θα γίνει στο Συμβούλιο και ελπίζω πριν από την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στο τέλος του τριμερού διαλόγου της 9ης του μηνός λάβαμε τη δέσμευση του Συμβουλίου ότι θα συμμετάσχει σε μια άλλη κοινή συνεδρίαση για τις πληρωμές που θα γίνει όμως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με... και αυτή τη φορά θα είναι παρόν εν πάση περιπτώσει του Συμβουλίου που είναι εκ των όνων κάνευ για να έχουμε μια κοινή βάση, για να έχουμε ένα κοινό σημείο θετήριας για τη συνδιαλλαγή. Από την άλλη, λάβαμε μια κοινή δήλωση γραπτή μάλιστα, που θα δούμε τι μορφή θα πάρει τις επόμενες ε, μέρες από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Giovanni. Σε ευχαριστούμε, Τζοβάνι. Ντέρεκ. Ντέρεκ Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ο κύριος ε, Λαβία νομίζω ότι παρουσίασε τη γενική θέση πολύ καλά. Ήμουν στον τριμερή διάλογο για να δω τα άλλα το... Ε, την κατηγορία 5. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος. Ως αποτέλεσμα έχουμε καλύτερες ιδέες για τον τρόπο σκέψης του Συμβουλίου για τον διοικητικό προϋπολογισμό των θεσμικών οργάνων. Λένε ότι θέλουν όλα τα θεσμικά όργανα εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παγώσουν στους προϋπολογισμούς και υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, δεν πήραξαν το δικό μας, αλλά για τα άλλα θεσμικά όργανα προτείνουν πάγωμα για το 2013 του προϋπολογισμού και αν περάσει η αύξηση από, από το 2,3% που θα πάει στο 1,4%. 1,47%. Το Συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε την αύξηση 1,7% στους μισθούς γιατί έγινε προσφυγή στο δικαστήριο. Μάλλον, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα χάσουν, οπότε θα δούμε ότι θα υπάρξει το 1,7%. Είπαμε στον τριμερή διάλογο να συμπεριληφθεί το 1,7% στον προϋπολογισμό τώρα, αφού έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουν στο μέλλον. Επίσης, ε, για τις άλλες κατηγορίες θα πρέπει να δούμε κάθε θεσμικό όργανο χωριστά, γιατί θα ήταν λάθος να παγώσουμε τα πάντα για κάθε θεσμικό όργανο που είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους και με διαφορετικές ανάγκες και χρειάζονται κάποιες αυξήσεις. Ε, δεν θέλουμε αυτή την οριζόντια περικοπή, αυτό το οριζόντιο πάγωμα. Πρέπει να δούμε χωριστά κάθε θεσμικό όργανο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και ως Επιτροπή Ευχαριστώ. Σαλβαδόρ Γκαρίδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτές ε, οι δηλώσεις ε, του Συμβουλίου σε μια τόσο πρώιμη στιγμή ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη συζήτηση του προϋπολογισμού τον Ιούλιο δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αυξήσει από ό,τι φαίνεται σημαντικά το 2,79 των πληρωμών. Αλλά αυτό ξέρετε είναι μια κακή πρακτική γιατί αν κάναμε και εμείς το ίδιο τότε θα έλυγε άμεσα η διαδικασία κατάρτισης του προπολογισμού και θα πηγαίναμε στα 12 τιμόρια. Δεν είναι καλός τρόπος να ξεκινά μια τέτοια διαδικασία κατάρτισης προπολογισμού. Αυτό δεν που δείχνει είναι μια πάρα πολύ κλειστή στρατηγική από το Συμβούλιο και όπως ε, είπε και ο εισηγητή, είναι και εντελώ αντιφατική η στάση σχέση με τι συμφωνίε οι οποίε είχαν ληφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη 29 η Ιουνίου. Ε, τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην θεωρήσουμε δεδομένη αυτή την δήλωση του Συμβουλίου για το 2,79% και να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, να συνεχίσουμε να ζητούμε πιο ε, πλήρες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο και ιδίως από το Συμβούλιο. Γιατί από την πλευρά της ε, Επιτροπής Υπερπολογισμού του Συμβουλίου πρέπει να δούμε τι βλέπουν ε, ότι θα υπάρχει ω επίπτωση με το 2,79 πιστός πλήρωμων. Δεν θα πειράσει αυτό τις ίδιες τις γραμμές του προπολογισμού τις οποίες κρίνει και έχει δηλώσει ότι είναι σημαντικές το ίδιο το Συμβούλιο για να έχουμε αυτό το σύμφωνο για την ανάπτυξη. Επειδή έχουμε και εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, εμένα θα με ενδιαφέρει και θα ήθελα να συζητήσουμε και ένα ε, ζήτημα που σε αυτή τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου για τι πληρωμέ πρέπει και να, να το θέσουμε αυτό το θέμα. Ε, άλλωστε, είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση ε, ούτω ή άλλω, γιατί αλλιώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να πάμε στη συνδιαλλαγή του Νοεμβρίου. Τώρα, ε, πράγματι υπάρχουν αρκετέ αντιπροσωπείε στο Συμβουλίου οι οποίε θεωρούν ότι η έλλειψη δέσμευση που βλέπουμε του τελευταίου μήνε ε, θα συνεχίσει να είναι μαζική. Και επομένω δεν χρειάζεται να αυξηθεί αυτό το ποσοστό των πληρωμών για το προσεχέ έτος, αυτό το 2,79%. Διότι ο διορθωτικό προπολογισμό που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιλαμβάνει επαρκή ε, χρήματα. Αυτή είναι μια θεωρία. Είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να, ε, να μας ενημερώσει σχετικά τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τέλη του έτους. Ε, διότι αν πράγματι δεν έχουμε εκτέλεση όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και για το 2,79, ε, όχι βέβαια αυτό το 6 και κάτι που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μας πει βασικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με τις αναλήψεις υποχρεώσεων Ευχαριστώ πολύ, για πρόταση, Έλκα Τρούπελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Πρέπει να πω ότι αυτό που πρότεινε τώρα το Συμβούλιο δεν είναι απρόβλεπτο, το περιμέναμε, αλλά είναι άσχημη η πρόταση. Συμφωνώ με τους εισηγητές και με τον Σαλβαντόρ Ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε τα νούμερα, την αύξηση στις πληρωμές μόνο 2,7% με τα νούμερα της Κομισιόν 6,8%. Όλοι ξέρουμε ότι στην πολιτική αντιπαράθεση, πολιτικό επίπεδο, το 6,8% φαίνεται πολύ ψηλό αλλά σε σύγκριση με την ανακοίνωση των κρατών μελών προς την Κομισιόν, τι θέλουν δηλαδή, ήταν πολύ μετριοπαθής η πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό πάντοτε ε, δικαιολόγησα την ε, πρόταση αύξησης της Κομισιόν. Τώρα βλέπουμε μια παραδοσιακή πολιτική προσέγγιση όπου το Συμβούλιο θέλει να περικόψει στην κατηγορία 1α πολιτικές ανάπτυξης, ε, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνισμός, σε βάρος ε, των πολιτικών μας προτάσεων. Είναι πολύ παράδοξη πολιτική κατάσταση αυτή. Είπε ο Σαλβαντόρ ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος δεν θα υπάρξει συμφωνία στον προϋπολογισμό του 2013. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα θα διαπραγματευτούμε τον προϋπολογισμό του 2013 και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο παράλληλα. Οπότε είναι σαφέστατο νομίζω ότι από άποψη στρατηγικής πρέπει να συνδυάσουμε τις δύο πολιτικές προκλήσεις γιατί αν είναι πολύ κακή η έκβαση από τον προϋπολογισμό του 2013 και συμφωνούσαμε σε αυτό, τότε θα διαμορφωνόταν δυσμενέστατη κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές και τα νούμερα που θα θέλαμε για τον προϋπολογισμό του 2013 και τη θέση μας που πέρασε με πάνω από τα 500 ψήφους, τα νούμερα δηλαδή του 2013 συν 5%. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε αν δεν υπάρχει πραγματικά, πραγματική βελτίωση, όπως είπε ο Σαλβαντόρ, να είμαστε έτοιμοι να πούμε όχι, γιατί είναι το μόνο μας όπλο ενάντια στο Συμβούλιο, για να έχουμε στεναρή θέση. Αν δεν είναι σαφές αυτό, ε, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με στεναρό τρόπο. Οπότε θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων επί της πολιτικής στρατηγικής μας και θέλω βέβαια να ξέρω τι θα πει και η Κομισιόν γιατί θα πρέπει να δούμε τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχουν τα νούμερα που έδωσε το Συμβούλιο. Από τη δική μας την άποψη και έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα τώρα, ρισκάρουμε να μειώσουμε τα ποσά για έρευνα και ανάπτυξη και για πολλά άλλα θέματα που θεωρούμε εμείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και από την άλλη πλευρά Ξέρω βέβαια ότι δεν συμφωνείτε, αλλά για παράδειγμα διατηρούμε την πρόταση του Συμβουλίου, με την πρόταση του Συμβουλίου τις πληρωμές για το Ίτρε αλλά θα μειώσουμε τις ε, πληρωμές για ερευνητικά προγράμματα και αυτό δεν μπορεί να είναι προς συμφέρον μας αν θέλουμε μια φιλόδοξη στρατηγική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν διατηρούμε το ίτερ, αλλά μειώνονται τα ερευνητικά. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η επαρκής ε, ε, βελτίωση και αν δεν είναι επαρκή και ικανοποιητική, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε όχι. Ευχαριστώ, Χέλγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκαρδία Θάμπαλ, Ρουμπιάλ. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα ε, συμφωνούμε με αυτά που υπόθηκαν. Ο τριμερής διάλογος της προάλλης δεν ήταν καθόλου παραγωγικός. Βέβαια ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Δεν ήθιστε να προχωρούν και πολύ τα πράγματα τον Ιούλιο. Τουλάχιστον συμφωνήσαμε να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή για αυτή τη γραπτή δήλωση. Τέλο πάντων, ε, πάντοτε δεσμεύονται ότι θα χρηματοδοτήσουν τα πάντα, ότι είναι απαραίτητο και μετά καταλήγουμε να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με το Συμβούλιο για αυτή τη χρηματοδότηση. Πάντω το Συμβούλιο δεσμεύτηκε ότι θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ και να μιλήσει για τι πληρωμέ και με το, Συμβούλιο, με το, συγγνώμη, με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει λοιπόν το Συμβούλιο μόνο αύξηση κατά 2,79 πληρωμέ. Τι περιθώρια αφήνει αυτό στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο. Κανένα ουσιαστικά. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε, ε, να βάλουμε το Συμβούλιο να ανοίξει τα χαρτιά του και να μας πει τι δεν θα χρηματοδοτήσει. Πάνω από πέντε δις, όχι ότι θα τα δεσμεύσουν, αλλά δεν θα τα δαπανίσουν για τις πληρωμές πού, από πού θα φύγουν αυτά τα χρήματα, τι δεν θα χρηματοδοτηθεί, ερευνητικά ε, προγράμματα, υποτροφίες, εράσμους, πανεπιστήμια, να μας πούν τι δεν θα χρηματοδοτήσουν. Και τι στρατηγική πρέπει να έχουμε, λέγει Χέλγκα. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε κάποια στρατηγική. Ε, νομίζω πρέπει να πούμε όχι, τελεία και παύλα, αυτό είναι το ένα, ή να πούμε, ωραία, θέλετε αυξήσετε μόνο κατά 2,79 πληρωμέ. Το δεχόμαστε αυτό το ποσοστό. Αλλά σε όλε τι γραμμέ, του προπολογισμού θα μπει αυτό, εκτός από τις γραμμές όπως τα ταμεία συνοχής, όπου τα χρήματα επιστρέφουν στα ταμεία των κρατών μελών. Σε πολλές χώρες θα γίνει πόλεμο στην Ισπανία, στη Γαλλία ίσως, αλλά ε, αυτοί φαίνεται ότι δεν θέλουν να βάλουν χρήματα. Ας μην δώσουν χρήματα, δεν θα πάρουν και χρήματα από αυτές τις κατηγορίες που προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων στις ε, χώρες μέλη. Είναι ένας παραλογισμός αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε με το Συμβούλιο. Όπως έλεγε ο Σαλβαδόρ, μπορεί να φτάσουμε και σε σημείο να μην γίνονται συνδιαλλαγή ούτε προπολογισμό. Αν υπάρξει αδιέξοδο στι διαπραγματεύσει. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια σοβαρή αντιμετώπιση. Γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να πούμε όχι και να τελειώνουμε ή να πούμε ναι, δεχόμαστε αυτέ τι περικοπέ, αλλά εμεί θα πούμε που θα γίνουν οι περικοπέ και αποκαθιστούμε την ε, γεωργία, την κατηγορία 1α, δηλαδή την 4 κτλ. κτλ. Δεν ξέρω ακριβώς τι στάση πρέπει να τηρήσουμε στην Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό που ακούμε ότι διαπαραταξιακά ε, υπάρχει ενότητα σε αυτά τα θέματα, γιατί η αντιμετώπιση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο και η αντίδρασή μας δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα θεσμικό και η συμπεριφορά του Συμβουλίου δείχνει ότι αργά αλλά σταθερά σε πολλούς τομείς προωθείται από ευρωπαϊκοποίηση του Συμβουλίου. Οι συνάδελφοι σε άλλε επιτροπέ θα το δουν και αυτοί στους τομείς τους. Εγώ το είδα στο Σένιεν, στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και το βλέπουμε και σε άλλα σημαντικά θέματα. Οπότε ήρθε η ώρα να στείλουμε ένα μήνυμα, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ε, κάνουμε προϋπολογισμό, λες και είναι ένα μικρό μάγαζο που μπορούμε να το προσαρμόζουμε όπως θέλουμε. Πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα. Το κάναμε άλλωστε επιτυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ συμφωνώ και υποστηρίζω τους δύο εισηγητές ε, σε αυτά τα θέματα. Και είναι και σωστό αυτό που είπε η συνάδελφος Τρίπελ για τη στρατηγική που πρέπει να τη σκεφτούμε εμείς για να δώσουμε καλές ε, προτάσεις. Πρέπει να συζητηθούν τα θέματα αυτά και με τους ε, σκιώδεις, ούτως ώστε η στρατηγική αυτή να είναι αποτελεσματική. Πολλές φορές ε, βλέπω ότι είναι ε, ε, μικρή η μνήμη του Κοινοβουλίου, βραχία μνήμη, γιατί ε, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να γνωρίζουν ότι πρέπει να δοθεί μήνυμα σωστό προς τους λαούς της Ευρώπης. Δεν μπορεί να δίνουμε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό θα είναι επιζήμιο και καθόλου αξιόπιστο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω την προσέγγιση του Συμβουλίου. Και οι προτεραιότητες που όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία, που εγκρίθηκαν ε, με συντριπτική πλειοψηφία, να ισχύσουν. Ε, βεβαίως είναι συνδεδεμένο το θέμα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και περιμένουμε ενδιαφέρον οδόν θα υπάρξει καλός διάλογος εδώ. Ιδιαίτερα όταν θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο οι διαπραγματεύσεις, δεν θα πρέπει να επικριθεί το Κοινοβούλιο ότι ε, δεν ανταποκρίθηκε στις ε, ανάγκες που έχουν οι διάφοροι πολιτικοί τομείς. Νομίζω ότι αν υπάρξει αποτυχία σε ορισμένους τομείς και χρειαστεί να μειωθούν οι πιστώσεις πληρωμών, σε σημαντικούς τομείς θα πρέπει να καταδειχθεί ο υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Σε συνεργασία με την Κομισιόν νομίζω ότι θα υποβληθεί ρεαλιστική πρόταση. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά να κάνουμε αυτά τα παζάρια για ένα αυτή τη κλίμακα ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Όπως και οι συνάδελφοι από τις άλλες ομάδες και εμείς θεωρούμε αξιολύπητη τη θέση και κατακριτέα τη θέση του Συμβουλίου. Ιδίως ό,τι αφορά αυτή την αύξηση του 2,79% των πληρωμών. Η Κομισιόν είχε προτείνει υψηλότερο νούμερο. Έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα μια φορά αυτή η πρόταση πλήττει το τα προγράμματα για την απασχόληση, για την ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα κτλ. Του συνήθεις υπόπτου. Είναι τα συνήθη θύματα. Είναι προγράμματα, όλα τα προγράμματα δηλαδή που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και αυτό έρχεται σε αντίφαση, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, με την ιδέα που προωθούν οι κυβερνήσει ότι θέλουμε δηλαδή περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι το Συμβούλιο γελιοποιείται με αυτή την πρόταση. Δεν συνειδητοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ε, θα συνειδητοποιήσουν αυτή τη γελιότητα της τάσης του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την πρόταση του 2,8% που είναι παντελώς ανεπαρκής. Βεβαίω ε, μπορούμε να κάνουμε διορθωτικούς προπολογισμού στο μέλλον, αλλά με αυτό το προπολογισμό ε, επιδεινώνουμε το πρόβλημα και δεν λύνουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια τώρα και από τη δική μου την πλευρά. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια μεγάλη ομοφωνία, μια μεγάλη συνένεση στην Επιτροπή Προπολογισμών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας, της 28ης και 29ης Ιουνίου, εισήγαγε δύο σημαντικά στοιχεία. Πήρε δύο σημαντικές αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2013. Η πρώτη απόφαση είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα που επιθυμεί για την υιοθέτηση του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και όλων των κανονισμών και των πολιτικών που χρηματοδοτεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Το χρονοδιάγραμμα είναι προθεσμίες. Η προθεσμία είναι Δεκέμβριος του 2012. Αυτό τι σημαίνει, ότι στην πράξη το χρονοδιάγραμμα διαπραγμάτευσης για τον προϋπολογισμό του 2013 και του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα ε, συμπέσουν κάπου. Και τον, ε, το φθινόπωρο θα δούμε πώς θα τα διευθετήσουμε αυτά, πώς θα τα καταφέρουμε, ξέροντας ότι η ψηφοφορία που μπορεί να γίνει για το ένα θέμα θα είναι μήνυμα για το άλλο θέμα. Θα είναι έτσι μια πρόγευση για το δεύτερο θέμα, το πολιετές δηλαδή πλαίσιο. Η δεύτερη απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η εξής. Παναλαμβάνω αυτό που είπαν οι συγκητές εδώ και κάποιοι ομιλητέ. Και είναι πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μία πολιτική δήλωση στο, με τίτλο «Σύμφωνο Ανάπτυξης». Αντίστοιχο με το Fiscal Compact. Σύμφωνο δηλαδή δημοσιονομικό. Το δεύτερο είναι μια συνθήκη. Ε, το άλλο, ε, το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη, είναι μια πολιτική δήλωση όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγγέλει και δηλώνει τη θέλησή του να δώσει 130 δις ευρώ επιπλέον για να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και δίνει και κάποιες λεπτομέρειες για την κατανομή αυτών των 130 δις, λέγοντας ότι αυτό θα πρέπει να σημαίνει Συμπληρωματικέ πιστώσει για την έρευνα, την καινοτομία και 55 δις επιπλέον για τα διαφορετικά ταμεία που θα πρέπει να αποκτήσουν νέο προσανατολισμό για προγράμματα πιο καλά υπέρ της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της γρήγορης ανάπτυξης μάλιστα. Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος την επαύριο της συνεδρίασης της, της Κομπιούτα που έγινε υπό την αιγύδα της Κυπριακής Προεδρίας του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών. Στον τριμμένο διάλογο διαπιστώσαμε ότι σε Συμβούλιο Υπουργών, σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, συγγνώμη, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν ελήφθη υπόψη καθόλου. Αγνοήθηκε παντελώς. Και αυτό μας κατέπληξε βέβαια. Το έκανα, ε, ξέφρασα αυτή την κατάπληξή μου σε ένα ανακοινοθέν. Και μαζί με τους συζητητές ε, τα είπαμε αυτά, αυτή, δηλώσαμε αυτή την κατάπληξη που αισθανόμαστε στον τύπο. Έθεσα το ερώτημα και στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι και στο Συμβούλιο για την ερμηνεία που δίνουν στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι σήμαινε αυτή η απόφαση είπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θέλει επιπλέον επιστώσεις και μάλιστα 55 δις επιπλέον για τα διαφορετικά ταμεία. Προσθέτοντας ότι στα πλαίσια ότι θα έχετε ακούσει κι εσείς όπως και εγώ από την Κομισιόν να μας λέει κατά διάρκεια της Ολομέλειας της, του Στρασβούργου, την Τρίτη όταν ήρθε και ο Φαν Ακούσαμε λοιπόν από πλευρά ε, διαστόματος Μπαρόζο να μας λέει η Κομισιόν ότι ήδη 20 δισεκατομμύρια ευρώ πιστώσεις για τα διαρθωτικά ταμεία έχουν επαναπροσανατολιστεί προς πιο ενδιαφέροντες προορισμούς. Και τα 55 δις που είχε αναγγείλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του θα προσθεθούν εκεί. Κατά τη διάρκεια όμως του τριμερούς διαλόγου Ούτε ο Κύπριος Υπουργό, ούτε ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι απάντησαν ή ήταν σε θέση να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αυτό το που τους κάναμε, ποια είναι η ερμηνεία που δίνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι 55 δις, είναι 20 δις, είναι πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων, είναι πιστώσεις πληρωμών, είναι ε, κατάλοιπα μη χρησιμοποιημένων πιστώσεων από πέρυσι που υπάρχουν στα ΡΑΛΣ, είναι προβλέψεις για την χρήση 2012, είναι πιστώσει για το 2012-2013, είναι επιπλέον πιστώσεις, αλλά προστίθενται σε τι. Τέλος όλες αυτές τις ερωτήσεις τις άφησαν αναπάντητες. Έγραψα λοιπόν μια επιστολή και εγώ, για να ζητήσω από τους υπουργού επίσημα γραπτά, τον Υπουργό της Κυπριακή Προεδρία και από τον Επίτροπο και να ρωτήσω και τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι τι έχουν να μας πούν, ούτω ώστε να ξέρουμε κι εμείς πώς να ερμηνεύσουμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό για μας όταν θα ψηφίσουμε για το σχέδιο προπολογισμού του 2013. Και το διορθωτικό προπολογισμό του 2014. Αυτά έγιναν τη Δευτέρα. Την Τετάρτη το πρωί, χθε, είχαμε το κορεπέρ. Ένα κορεπέρ εντυπωσιακό Καταρχάς, όπως είπε και η Χέλγκα Τρούπελ, το αποτέλεσμα δεν ήταν ε, εντυπωσιακό, δεν ήταν κάτι που δεν περιμέναμε, αλλά πάντως δεν ήταν και καλό. Επιβεβαίωσαν αυτά που είχε πει η Κομπιτ. Ούτως ή άλλως τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, βάζουν σφραγίδες σε αυτά που λένε οι υπάλληλοι του προϋπολογισμού. Εκεί που γίνεται το πράγμα ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υιοθέτησαν μία πολιτική δήλωση για τις, για τις πληρωμές. Η πλειοψηφία που ψήφισε το σχέδιο προπολογισμού είναι ειδική πλειοψηφία, δεν είναι ομοφωνία. Και υιοθέτησε μία δήλωση για τις πιστώσεις πληρωμών. Υιοθετήθηκε από όλε τι αντιπροσωπείε εκτό από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Σουηδία και τι κάτω χώρε που ψήφισαν κατά του σχεδίου προπολογισμού. Οκ. Και η Αυστρία που απήχε. Οι πόλοι ψήφισαν το σχέδιο προπολογισμού και τη δήλωση. Να σα διαβάσω τη δήλωση. Το Συμβούλιο ζητάει από την Κομισιόν να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν το, την επιστολή τροποποίησης για τη γεωργία και τις πληροφορίες για τις μεταφορές και αν χρειάζεται μία επιστολή για την κατηγορία 1β, ούτω ώστε να υπολογίσουμε το επίπεδο των πόρων στο, στην κατηγορία 2 και στην υποκατηγορία 1β στον προϋπολογισμό του 2013. Επιπλέον, το Συμβούλιο ζητάει από την Κομισιό να υποβάλει ε, ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, γιατί ο προϋπολογισμός του 2012 είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες του 1α και 1β, του, της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 4. Καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ε, νέα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση των πραγμάτων και τις εκτιμήσεις ό,τι αφορά τις πιστώσεις ε, αναλήψης προμών στην ε, υποκατηγορία 1β και αν χρειαστεί ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού με μόνο σκοπό να λάβει θέση το Συμβούλιο ε, στο σχέδιο προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, τόσο ώστε να μην έχουμε λήψεις στις α, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Καλά νέα. Λοιπόν, το Κορεπέρ γνώριζε τι θέληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνει κάτι για τις πληρωμές. Αλλά Εφτά χώρες, οι τέσσερι που δεν ψήφισαν υπέρ τη δήλωση. Και που είναι λογικό. Αλλά και ακόμα τρεις χώρες που ψήφισαν υπέρ τη δήλωση. Που ήταν η Γαλλία, η Γερμανία και η Φιλανδία. Υιοθέτησαν επίσης την εξή δήλωση. Αναφέρω. Δημοσιονομική, η δημοσιονομική λιτότητα και οι περιορισμοί ε, σε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική προκειμένου να διορθώσουμε τα δημόσια οικονομικά μας για να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Ε, η αύξηση 2,79% είναι υψηλότερη από αυτό που θα θέλαμε. Επομένως, περαιτέρω αυξήσεις στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να συμφωνηθούν αργότερα μέσα στο 2012. Είναι παλαβό. Είναι παλαβό. ίδιες χώρες δηλαδή. Την ίδια μέρα για το ίδιο θέμα τη ημερήσιας διάταξη, Από τη μία λένε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, προσοχή, προσοχή. Γιατί αν λείψουν οι πιστώσει, πληρωμών φέτος, θα πρέπει να μας κάνετε προτάσεις για να τις βρούμε αυτέ τις πιστώσεις, για να, να αυξήσουμε τα χρήματα. Και αμέσω μετά λένε, α, κάναμε πολλές ε, μειώσεις, πολλές περικοπές στο σχέδιο προπολογισμού του επόμενου έτου, αλλά θέλαμε περισσότερε περικοπέ. Αυτό ο προπολογισμό είναι πολύ γενναιόδωρος και σας λέμε ότι ό,τι και αν συμβεί δεν πρόκειται να σα δώσουμε ούτε δεκάρα μέσα σε όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω εσεί πώ αντιδράτε σε αυτά. Εγώ προσωπικά έχω την πρόθεση να δημοσιεύσω την εξής, το εξής ανακοινοθέν. Προσωπικό είναι και δεν θέλω να σας ανησυχήσω. Διαβάζω το δημοσιονομικό πρόβλημα σε σχέση λοιπόν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την κρίση του χρέους και τον ε, προϋπολογισμό, ε, θα σας τα διαβάσω στα γαλλικά αργά αυτά τα οποία θέλω να πω. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ήδη είναι άκρος Ωστόσο, τα μειονεκτήματά της επιδεινώνονται πλέον από λόγω μάλλον ε, περίεργων δυσλειτουργιών σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κρίθηκαν ομόφωνα. Ωστόσο, <clears throat> το περιεχόμενο της συμφωνίας ε, στο άκρος ε, υψηλό επίπεδο δεσμεύει μόνο, ε, μάλλον δεν δεσμεύει καθόλου τις κυβερνήσεις που τελικά το αμφισβήτησαν το κείμενο αυτό δύο μετά. Δύο συγκεκριμένα χώρες και μια τρίτη χώρα η οποία ε, επιλήφθηκε το θέμα του συνταγματικού δικαστήριο αναβάλλοντα για το φθινόπωρο την απόφαση. Το εμβληματικό σημείο ήταν η ανάπτυξη ε, στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξη που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Κυπριακή Προεδρία των, ε, του Συμβουλίου Υπουργών εξέφρασε την ικανοποίησή της που αυτό μεταφράστηκε σε μαζική μείωση των κονδυλίων για την έρευνα, την καινοτομία και τη συνοχή που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013. Για λόγους πολιτικής ευγένειας θα μπει στον λογαριασμό των πρέσβεων το γεγονός ότι τρεις, δηλαδή ο Γερμανός, ο Φιλανδός και ο Γάλλος, την ψήφο τους για τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό την συνόδευσαν με δύο δηλώσει τελείω αντιφατικέ μεταξύ τους. Η πρώτη καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει γρήγορα αιτήματα για ε, πρόσθετες πιστώσεις εκεί που θα φαίνονταν ότι ήταν περικοπέ περικοπές προπολογισμού. και η δεύτερη δήλωση που την υπογράφουν οι ίδιοι ακριβώς εκφράστηκε τη λύπη τη ε, για το ότι ήταν ανεπαρκείς οι περικοπές και ανακοινώνει ότι αυτές οι χώρες ε, θα αρνηθούν οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματοδότηση. Υπάρχει λοιπόν ε, πλήρης ασυνέπεια και ανευθυνότητα η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο, σε σοβαρό κίνδυνο την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα σημείο χρονικό όπου αυτό θα ήταν άκρος απαραίτητο να υπάρχει, αξιοπιστία δηλαδή. Δεν από το εγκόμιο βέβαια όπως καταλαβαίνετε. Δεν σας προτείνω να το προσυπογράψετε, Αυτά θα τα πω πάντως εγώ και αν κάποια από εσάς θέλετε να εκφράσετε συγκρίσιμα παρόμοια σκέψεις και συναισθήματα να το κάνετε γιατί πρέπει να τα λέμε, πρέπει να μιλήσουμε πλέον. Έτσι λοιπόν συνάδελφοι, για το σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Θα ζητήσω λοιπόν από τον Τζοβάνι να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Μετά από όλη αυτή την ε, γλαφυρή παρουσίαση του Προέδρου Λαμασούρ, ας πάμε στο, πάλι στο χάος του Συμβουλίου, όπου η αριστερά δεν γνωρίζει τι πει η δεξιά. Και η αριστερά λίγες πολύ σύντομα, χρονικά, κάνει δύο αντιφατικές δράσεις ε, μεταξύ τους. Επανέρχομαι τώρα στον προπολογισμό και στα πιλωτικά προγράμματα. Όπως θα θυμάστε, παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο αρχές Ιουνίου όλες τις προτάσεις μας για τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις και τις στείλαμε στην Κομισιόν, ούτω ώστε να κάνει μια αρχική αξιολόγηση για την σκοπιμότητα πριν συνεχίσουμε τη διαδικασία του προϋπολογισμού και έγκαιρα, ούτω ώστε να κάνει και κάποιες προσαρμογές, αν θέλει. Ούτω ώστε να είναι εύκολα εφαρμόσιμες αυτές οι προτάσεις του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε επίσης, το Κοινοβούλιο είχε παρουσιάσει ένα κατάλογο από 142 προτάσεις, πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις, της απίφθηνες στην Κομισιόν, για να τις αξιολογήσει. Συνολικά αυτές οι προτάσεις έφταναν στα 232,7 εκατομμύρια ευρώ ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και θα θυμάστε ότι το όριο των πιστώσεων υποχρεώσεων για τα πιλωτικά προγράμματα στον υπολογισμό είναι ίσο με 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συνήθως, έκανε την αξιολόγηση σκοπιμότητας και ε, κατηγοριοποίησε τα προγράμματα ε, σε τέσσερις κατηγορίες. Και από τις 142 προτάσεις ε, που δώσαμε, μας επιστρέφει 29 ε, της κατηγορίας Α, δηλαδή που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τροπολογίες, χωρίς το τροποποίησης. 19 μπορούν να εφαρμοστούν μερικά ή πλήρως με κάποιες αναθεωρήσεις και επομένως χαρακτηρίζονται στην κατηγορία Β 73 προτάσεις που, προβλέπει το Κοινοβούλιο καλύπτονται από νομική βάση και 17 δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχουμε και τέσσερα προτάσεις ακόμα, για τις οποίες δεν έχουμε λάβει απάντηση από την Κομισιόν και περιμένουμε. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση της Κομισιόν μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα πρέπει βεβαίως στη συνέχεια της διαδικασίας να αξιολογήσουμε τις προτάσεις και το ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις μπαίνουν ε, στην κατηγορία 1α. Από τις 50, 51 από τις 142 ε, μπαίνουν στην 1α. Και στο σχέδιο προπολογισμού είχαμε ένα περιθώριο 91 εκατομμύρια ευρώ. 19 προγράμματα αφορούν την κατηγορία 3β και σε αυτή την περίπτωση το περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι προτάσεις με βάση την αξιολόγηση της Κομισιόν και αυτοί που προτείνουν αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ξαναδούν τις προτάσεις τους για να κάνουν αλλαγές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της διαδικασίας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το περιθώριο που έχουμε στην κάθε κατηγορία ε, στην τελική πρόταση που θα κάνουμε για τις ε, ε, τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Κάτι ακόμα που μου φαίνεται σημαντικό και πρέπει να τονιστεί. Αυτή η προκαταρτική αξιολόγηση της Κομισιόν μας δίνει ένα νέο στοιχείο για να κάνουμε και εμείς αξιολόγηση των δικών μας προτάσεων και μπορεί να μας επιτρέψει να τις βελτιώσουμε, τις προτάσεις μας. Τώρα, θα ξαναδώσω το λόγο του, στα άτομα που προτείνουν αυτά τα προγράμματα, μήπως πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές και με βάση και τη θέση της Κομισιόν ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια ιεράρχηση των προτάσεων αυτών, ούτω ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια της τελικής συμφωνίας να κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση και να έχουμε ένα πακέτο προγραμμάτων, έργων και project που θα ε, εφαρμοστεί στην επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας προτείνω να εμβαθύνουμε λίγο στο περιεχόμενο και στην εμβέλεια ενός πολύ σημαντικού, όπως και όλων, ε, πιλωτικού προγράμματος. Ε, ο συνάδελφος James Ellis θα μας πει σχετικά. Σε αυτό συμμετέχουν όλες τις μικρόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Jean-Claude που τον γνωρίζουμε πολύ καλά, ο Γενικός Διευθυντής ε, της είναι εδώ. Ο φίλος μας, ε, Μαρσίες Ποπόφσκι, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΙΕΔ, επίσης είναι εδώ και ο κύριος Μάτιου ο οποίος ανήκει στη γάμα πολιτικά θέματα του Συμβουλίου. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι όλοι σας, διότι θα πρέπει να περάσουμε ευθύς αμέσως στην ε, ψηφοφορία. Αλλά πρώτα να δώσω το λόγο βέβαια στον James Ellis. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να είμαστε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, πολύ ακριβείς. Εδώ μιλάμε για πρόθεση στρατηγικής προβλεπτικής σκέψης Πρέπει λοιπόν σύντομα να πούμε πώς συμμετείχαμε στο Κοινοβούλιο και να ακούσαμε και από τα άλλα θεσμικά όργανα πώς θα συνδράμουν όλα μαζί για να δημιουργηθεί στρατηγική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από άποψη Κοινοβουλίου μου, παρα... μου, ζητήσατε να παρακολουθήσω τις ε, πρωτοβουλίες ως συντάκτης της γνωμοδότησης. Έχουμε τρία στάδια. Πρώτα το πιλωτικό στάδιο που οδήγησε στο έγγραφο που έχετε μπροστά σας και που είναι πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Ε, έχει πολλά στοιχεία, ιδιαίτερα ε, την εξέλιξη των μεσαίων στρωμάτων, την καταναλωτική δύναμη μέχρι το, το, το 2013. Ε, πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας την εξέλιξη ψηφιακών υποδομών κλπ πριν ε, σκεφτούμε τον προϋπολογισμό του 2020 και υπάρχει και ένας άλλος βαθύτερος σκοπός που είναι στην παρασκευαστική δράση που εξελίσσεται τώρα για να εμβαθύνουμε την συγκέντρωση δικτύων ανώτερων αξιωματούχων που εργάζονται στα διάφορα θεσμικά όργανα για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ε, θα πρέπει να έχουμε απόλυτα λειτουργική ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό σύστημα ανάλυσης της στρατηγικής μέχρι το τέλος του 2014. Και για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας που θα δημιουργηθούν να δούμε την κοινωνία, τη διακυβέρνηση, να ε, έχουμε πραγματογνωμοσύνη εσωτερικά και εξωτερικά, δικτύωση σε μαζί με εκείνους που εργάζονται ε, στην Κίνα, στη Βραζιλία και αλλού, ούτω ώστε να μην μείνουμε στις Βρυξέλλες, να καταλάβουμε ότι γύρω μας ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Ε, έχουμε και ένα εστιακό τόπο που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την ταχύτητα των εξελίξεων έχετε αναφέρει ε, και εσείς ε, τρεις ε, ε, ανθρώπους που μπορούν να δώσουν τη μαρτυρία τους σε σχέση με τις εξελίξεις. ελπίζω να είναι όλα αυτά θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, James. Πράγματι, μας διανεμήθηκε αυτό το πρώτο έγγραφο που εκπώνησε αυτό το Think Tank. Δεν έχω βέβαια βρει χρόνο να το διαβάσω. Το Φιλομέτρησα όμως λιγάκι και το βρίσκω ενδιαφέρον. Κύριε Τιμπό, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να σας μιλήσω για αυτό το πραγματικά το project που δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά αν δεν είχε λάβει τη σχετική πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο James Ellis βέβαια όλος ιδιαίτερος ο οποίος ε, πρότεινε αυτό το πρόγραμμα και το οποίο εσείς υποστηρίξατε. Θα ήθελα λοιπόν ε, στο κοινοβούλιο σας να εκφράσω την ε, αμέριστη γνωμοσύνη όλων μας για την πρωτοβουλία αυτή που έχει προχωρήσει μέσω του πιλωτικού προγράμματος και βέβαια μετά με την προπαρασκευαστική δράση που ήδη είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είναι ένα σημαντικό project και θα σας πω για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα είναι καινοτόμο, είναι νεωτερικό και έρχεται να συμπληρώσει και ένα κενό. Ένα κενό που συνέσταται στο εξή. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, στρατηγικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν ένα εργαλείο ε, βοήθεια σε μια ε, διαδικασία λήψη ολοκληρωμένων στρατηγικών αποφάσεων. Έχουμε το National Intelligence Council τη ΕΠΑ ε, που καταθέτει στο γραφείο του κάθε εκλεγέντο Αμερικανού Προέδρου τι επιλογέ του. Αυτό δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιε εργασίε, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται κάτι τέτοιο για πρώτη φορά. Και βέβαια να προσθέσω ότι η κρίση δείχνει ότι αν ίσω είχαμε αναπτύξει μεγαλύτερη δυνατότητα και ικανότητα ανάλυσης και προοπτικής μελέτης, ίσως να ήμασταν πιο διορατικοί κατά το παρελθόν. Επίσης, άκρος πρωτότυπο είναι το διοργανικό ε, στοιχείο, διοργανικός χαρακτήρας αυτού του think tank. Υπάρχει με task force, στην οποία συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς των θεσμικών οργάνων, πολύ συχνά παρίσταται ο James Ellis, καθώς και υποφαινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αξιοσήμαντο και αυτό. Και τέλος είναι ένα project που δεν είναι, θα έλεγα, ευρωκεντρικό. Φυσικά και έχει δημιουργηθεί για να βοηθάει μας τους Ευρωπαίους, αλλά έχει να κάνει με τις ε, παγκόσμιες τάσει. Αυτές ε, εξετάζει. Και επομένως εργαζόμαστε με ανοιχτό πνεύμα ε, προτείνουμε ους. Υπάρχουν βέβαια κάποιες φορές ε, αντιφάσεις ίσως μεταξύ των ε, εταίρων ή των χαρακτών πολιτικής, αλλά και αυτό συνεισφέρει σε πλούσιες ε, συζητήσεις. Οδήγησε και στο πρώτο μας πόνημα το οποίο σας διανεμήθηκε και είναι ένα καλό έγγραφο. Σίγουρα επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση. Αυτό άλλωστε είναι και το αντικείμενο της προπαρασκευαστικής δράσης που έχει διδρομολογηθεί. Αυτή η προπαρασκευαστική δράση έχει ως στόχο κατά κάποιο τρόπο να εμπλουτίσει, να αναπτύξει τις εργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη πάντοτε με άνοιγμα προς τα έξω και με μία επικοδομητική αντιπαράθεση ιδεών. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι στο τέλος της όλης αυτής διαδικασίας ε, θα έχουμε ένα προϊόν, μια γενική έκθεση για τις τάσεις ε, με ορίζοντα το 2030, θα υπάρχει έπειτα και μια πιο πολιτική, ε, λειτουργική, επιχειρησιακή έκθεση, όπως θέλετε πείτε την, η οποία θα απευθύνεται στους προέδρους ε, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για την περίοδο 2014-2019. Και θα δούμε. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα προσλάβει ένα μόνιμο χαρακτήρα το project αυτό. Φυσικά και θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα άλλα ε, όργανα και να πω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία στο πλαίσιο της Task Force που θα συνεδριάσει μάλιστα σήμερα για μια ακόμη φορά και η οποία διαχειρίζεται καθημερινά το όλο project. Να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Γενικό της Γραμματέα τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, ο οποίο πραγματικά έχει δείξει μια μεγάλη δέσμευση προς αυτό το project. Να ευχαριστήσω και όλη του την ομάδα βέβαια. Η συνεχή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προφανές πως για μας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Να είστε πάντως βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτού του project Δουσουπουέ θα κάνει ό,τι μπορεί για να στεφθεί μέσω αίσιο πέρα σε αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις ε, φιλοφρονίες σας προς τον εισηγητή και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ποπόφσκι τώρα θα μας ε, πει την άποψη της τη της Ευρωπαϊκής, Επιτροπή, Εξωτερικής Δράσης και ίσως και κάποια πράγματα για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μας για τον ηγετικό ρόλο που έπαιξε το Κοινοβούλιο σας στο θέμα αυτό και το ρόλο του κυρίου Έλλης είναι πραγματική προσπάθεια ανάπτυξης μιας κουλτούρας στρατηγικής σκέψης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διοργανικός χαρακτήρας του εγχειρήματο είναι κέριος γιατί χρειάζεται η διοργανική προσέγγιση. Η πρώτη έκθεση ΕΣΠΑΣ λοιπόν ήταν μια επιτυχία, οπότε καλό είναι να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση και να ενισχύσουμε το κοινό έργο και, το, και η υπηρεσία εξωτερική δράσης ε, βεβαίως ε, ε, υποστηρίζουν. Υπάρχει προστιθέμενη αξία για τους εμπλεκομένους, ο προσανατολίζεται στην πολιτική, δημιουργεί υψηλής ποιότητας έρευνας. Βεβαίως είμαστε ρεαλιστές. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα βάση αυτό το πρόγραμμα για να αξιολογήσουμε την ωφελημότητα, την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων στρατηγικών πλαισίων, ιδιαίτερα στις εξωτερικές σχέσεις, όπως μακροπρόθεσμο πρίσμα για την ανάπτυξη των οργανισμών, ε, στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ε, που θα στρατηγική για την ε, ασφάλεια στο μέλλον. Το Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών της Ευρώπης συμμετείχε στη μελέτη και θα συνεχίσει να το κάνει. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι ο νέος διευθυντής του θα ε, διοριστεί σύντομα. Θέλω να επανεπιβεβαιώσω τη δέσμευσή μας λοιπόν και τη δέσμευση του Ιδρύματος του Ινστιτούτου αυτού που θα συνεχιστούν μια και έχω το λόγο και αν συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τον προϋπολογισμό της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η Κορεπέρα αρνήθηκε αύξηση για τον προϋπολογισμό. Συμφωνώ με τον κύριο Βον που παρατήρησε ότι πρέπει να δούμε μονομένα τα, τις υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα οι περικοπές δεν θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να λειτουργούμε του χρόνου και όπως το 2012. Ξέρουμε τι, τους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς ε, περιορισμούς και όπου μπορούν γίνονται. Όμως είμαστε στην πρώτη φάση και έχουμε ιδιαίτερες ανάγκες. Ε, ε, έχουμε 141 αντιπροσωπείες που αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών σε τρίτες χώρες. Επίσης αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του αδύναμου ευρώ και έχουμε πρόβλημα ασφάλειας της αντιπροσωπής στο Ιράκ, για παράδειγμα, ή το Αφγανιστάν. Ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση για την υποστήριξή σας, την υποστήριξη της Επιτροπής ε, υπέρ της ε, διαδικασίας του προϋπολογισμού συγκεκριμένα για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ φίλε. Ο εισηγητής μας σημείωσα την τελευταία παρατήρηση, ειδικά που ήταν πολύ σημαντική. Ο κ. Μάθιου Ρίτζ, από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ε, στις ευχαριστίες προς το Κοινοβούλιο και τον James Ellis για το πρόγραμμα αυτό. Όπως αναφέρθηκε, όντως υπάρχει ένα έλλειμμα ε, οι βασικοί μας εταίροι έχουν προχωρήσει ε, περισσότερο από εμά. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε και νομίζω ότι το κάναμε. Αυτό είναι το μυστικό. Το σημείο κινήσεως είναι ότι είναι καλό ότι τα θεσμικά όργανα προσανατολίζονται στο μέλλον. Είναι πολύ καλό να το κάνουμε αυτό όλοι μαζί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ευθυγραμμίσουμε τα καλύτερα στοιχεία που έχουμε στα θεσμικά όργανα με τα καλύτερα στοιχεία που μπορούμε να βρούμε εκτός θεσμικών οργάνων, είτε είναι αυτά think tanks ή συνεργασία με τους εταίρους και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα τελικό προϊόν που θα λαμβάνει υπόψη πώς διατέμνονται αυτές οι παγκόσμιες ε, τάσεις με τις πολιτικές και προκλήσεις της Ένωσης ε, για το επόμενο διάστημα 2014-2019. Αν φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε ένα προϊόν καλό, τότε θα έρθει μια στιγμή που θα απορούμε πώς είναι δυνατόν να μην είχαμε πάντα ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα ενδιαφέρονται για αυτή τη δουλειά. Συμμετέχουν ενεργά. Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Και όπως υπόθηκε, ο Κλάους Βέλε, ο Γενικός Γραμματέας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το τομέα. Και μάλιστα θέλουμε, θέλει να βελτιώσουμε την ικανότητα του Κοινοβουλίου να προβλέπει μακροπρόθεσμες προβλέψεις, να λαμβάνει υπόψη όλες τις εξελίξεις σε όλα τα θεσμικά όργανα. Πριν από δύο μέρες πήγε στο Παρίσι, στον ΟΑΣΕ, για να συναντήσει το Γενικό Διευθυντή του ΟΣΑ, συγγνώμη, για να δει πόσοι οικονομολόγοι που δουλεύουν στον ΟΣΑ μπορούν να συνεισφέρουν στο δικό μας οικονομικό προβληματισμό. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Σας προτείνω τότε να κλείσουμε αυτό το σημείο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη δυσκολία που έχουμε με τον ε, προϋπολογισμό του 2013 και θα επανέλθουμε και σήμερα το απόγευμα με την ε, εξέταση των οργανισμών, των agencies. Με βάση λοιπόν τώρα τη μέσια διάταξή μας, θα περάσουμε στις ψηφοφορίες ε, και μάλιστα θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Σας προτείνω να, να πάρετε αναχείρα τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Voilà, tout le monde a sa carte. Έχετε όλοι τι κάρτε σα. Σα παρακαλώ, λίγη ησυχία. Όσοι βγαίνουν από την αίθουσα να το κάνουν ησυχά ήσυχα. Θα ξεκινήσουμε. με το σημείο 21 και 22. Τις δύο εκθέσεις του κυρίου Κοσλόφσκι. Καταρχάς την έκθεση για το μέσο συνεργασίας με την πυρηνική ασφάλεια. Έχετε όλη την, τον κατάλογο ψηφοφορίας και το ΕΛΚΑ ακόμα. Πολύ ωραία. Πρώτο άρθρο. Τροπολογία 19. Helga Τσούπελ. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχέ. Απορρίπτεται. 20. Γκάιερ. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Δύο άτομα δεν ψήφισαν ακόμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δώδεκα υπέρ, 13 κατά, καμία αποχή. Ο Σαλβατόρε τρώει φιστίκια. Τι ψήφισες, παιδί μου. Κατά. Ο συντονίστης ξέχασε να ψηφίσει. 14 κατά, 12 υπέρ, απορρίπτεται. 8 του εισηγητή, υπέρ. Κατά. Άποχες. Υιοθετείτε. 21. 21 αποσύρεται. 22. Του κύριου Μουνίθ. Της κυρίας της κυρίας. Συγγνώμη κυρία μου. Η γραμματεία μπερδεύει τα φύλλα εδώ πέρα, δεν είναι σωστό. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννιά του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν. Υιοθετείτε. 23. Νιέσκι. Υπέρ είναι ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές υιοθετείτε. 10. Του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές είναι κατά. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Μιλάμε για την τροπολογία 10 του εισηγητή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ψηφίσουν, να ψήφισουν 27, αλλά ψήφισαν 26. Α, Σαλβατόρη, 28 με σένα. 27, πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 13 κατά, καμία αποχή. Σαλβατόρη, έχεις την κάρτα σου. 5 15 υπέρ, 13 κατά υιοθετείται. 11 του εισηγητή, που είναι συμβατή με την επόμενη. Υπέρ, κατά. Δύο εποχές. Καμία εποχή. Υιοθετείται. 24. που είναι συμβατή με την 11 που μόλις υιοθετήσαμε, αλλά το δεύτερο τμήμα Αποσύρεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 12. Που είναι συμβατή με την επόμενη. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ή μάλλον είναι του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε. 25. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 26. Γκάιερ. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. της Χέλγκα. Καταπίπτει γιατί υιοθετήσαμε τη 12. 13 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 28 της Μαρία Μουνή. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 29. Τρούπελ που συνάδει με την 28. Αλλά ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Μουνίθ. Υπέρ είναι ο εισηγητής. Ποιος, είναι υπέρ από εσά. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 31. Μουνίθ. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απέχουν οι φιλελεύθεροι. Υιοθετείτε. Όχι. Απορρίπτεται. Ας το τσεκάρουμε. Μιλάμε για την 31, ε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 31 της κυρίας Μουνίθ. Υπάρχει ένας από το, από το Λαϊκό Κόμμα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αποτέλεσμα. 15 κατά, 11 υπέρ, 5 εποχές απορρίπτεται. 32 τρούπελ. Ζήτης να κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 τρίπελ, ίδια κατάσταση, ο συγητής είναι κατά, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 34 της Χέλγκα. Σε τμήματα το ψηφίζουμε. Πρώτο τμήμα. Διαγραφή μέχρι το if appropriate supported. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Χέλγα. Και η Ιζαμπέλ. Ο Ζαν Λουκ διστάζει. Όμως κέρδισε η πολιτική πίστη σε σχέση με την εκτίμηση που έχουμε για τους συντάκτες. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Μία αποχή απορρίπτεται με πολύ κακό τρόπο. Το δεύτερο τμήμα, επομένως, θα πρέπει να ψηφιστεί τελικά. Deletion του τελευταίου, ε, deletion, του τελευταίου τμήματος. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οι περισσότεροι βέβαια. Αποχέ, αποχή απορρίπτεται. Δεν είναι τίποτα από την τροπολογία 34 της Χέλγκα. Αιτιολογικές σκέψεις. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, τις 3, 4 και 5 που είναι του συγητή, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετούνται και οι τρεις. 16 της Έλγα. Ο συγητήσαν είναι κατά. Υπέρ. Σοσιαλιστές και πράσινοι. Κατά. Οι υπόλοιποι. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 της Έλγα. Ο συγητήσαν είναι κατά. Υπέρ. η ίδια και η κυρία Βέρτμαν. Κατά. Απορρίπτεται. έξι της εισηγήτρια, του εισηγήτη, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 18. Μαρία Μουνίθ. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Πω, πω. Κοντά είστε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε ακόμα. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 14 κατά, συν ένα όμως που προσθέτουμε καμία αποχή. Wow. Je ne sais pas si on peut admettre un vote qui n'est que manuel, mais bon. Donc, il est rejeté. Κατά. Αποχές. Δύο Για την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Τοπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Δύο του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 14. Που είναι συμβατή της Μαρίας Μουνίθ. Ο εισηγητής είναι κατά μου. Είναι υπέρ. Αλλάζουν γνώμη ακόμη και ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι κατά. αποχές Υιοθετείτε. 15 που είναι συμβατή με τις προηγούμενες. Ο εισηγητής είναι κατά και εξακολουθεί να είναι κατά. Ο συντονιστής διστάζει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ζωζέ ψηφίζουμε. Το τελικό κείμενο. Le vote est clos. 26 plus 1, 27 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Υιοθετείτε. Συγχαρητήρια, κύριε Κοσλόφσκι που δεν είναι καν εδώ. Α, κοίταζα αλλού, μπροστά μου, αντί να κοιτάω αλλού. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια Γιάν. Συνεχίζουμε με σένα ούτως ή άλλως. Και τώρα έχουμε το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Έχετε όλο τον κατάλογο. Λοιπόν, το 8, εισηγή του υπέρ, κατά, αποχές υπέρ, εγκρίνεται περισσότερη. Σαράντα 45. Τι διαβάζω εδώ, ότι υπάρχει προφορική τροπολογία υπερθυμών 3 της κυρίας Brandner. out of budget scope. Υπάρχει κάτι που είναι εκτός του πεδίου, τέλος πάντων. Υπέρ η αριστερά. Κατά η δεξιά. Αποχές το κέντρο. Ας το ελέγξουμε τεχνικά, αστιαβόμουν, αστιαβόμουν. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά τροπολογία 45 εκτός του πεδίου της μετροπής. Μπάτσου. 13 ψηφιπέρ, 16 κατά, 5 εποχές. Απορρίπτεται. Α, έχετε την κάρτα σας, μάλιστα. Τέλος πάντων, ούτως ή απορρίπτεται. Πάμε στην 46 της κυρίας Μπραντνερ, προφορική τροπολογία πάλι εδώ, για να προσθεθούν οι λέξεις relevant indicators including. Κατά είναι ο εισηγητής. Ψήφι Κατά. Αποχή και μάλλον είναι αμφίροπο, γι' αυτό ηλεκτρονικά παρακαλώ να ψηφίσουμε. Άρχη ψηφοφορία. Είμαστε 33 και όλοι έχουμε την κάρτα μας πλέον, ωραία, οπότε. 17 υπέρ, 15 κατά καμία αποχή. Εγκρίνεται 46. 47 Μαρία Μουνίφρο, εισηγητής αντίθετος. 47, 48, 49. Μπορούμε μήπως να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι, δεν μπορούμε. Κρίμα. 47. Είναι αντίθετος εισηγητής. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. της αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η διαπεψηφία εγκρίνεται. 49 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή. Πάμε στην εννέα τροπολογία του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε, νομίζω είναι ε, περισσότεροι υπέρ, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, έρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 16 υπέρ, 10 κατά 6 αποχές, πράγματι εγκρίνεται. Τώρα, πού πάμε. Τροπολογία 10 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 Μπραντνερ είναι συμβατή. Κατά ο εισηγητής. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 του εισηγητή υπέρ κατά 2 αποχές ελεύθερη ναι, ναι, ναι. εγκρίνεται 51 είναι συμβατή της κυρίας Νιένης και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 του εισηγητή ψήφι υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 52 είναι ένισχυ και αυτή συμβατή ψήφι υπέρ. Κατά 2. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 ανιένσκι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 με μια προφορική τροπολογία. Ο εισηγητής υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αποχές εγκρίνεται. 55 της ιδίας ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 13 της ηγητή υπέρ κατά 3, 4, 5, 6, 7 αποχές 1 εγκρίνεται 56 Μαρία Μουνή, εισηγητής αντίθετος ψήφι υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 του εισηγητού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές προτιμώ να ελέγξουμε. 14 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλο και πιο πολύ γινόμαστε. Αλλά είναι πολύ παραπάνω συντηρητική από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ 14 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Η 14. Περνάμε στη 15 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα υποβάλω και τη 15 σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, αν και νομίζω την ίδια ψηφοφορία, αλλά Μιλάμε για μία με δύο ψήφου διαφορά, οπότε προτιμώ να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 17 κατά. Απορρίπτεται αυτή τη φορά και με μία αποχή. Εγκρίθηκε 14, απορρίφθηκε 15. Πάμε στη 16 η Δεν ψηφίζει το ΕΛΚ πια βλέπω. Ξέρετε, αρκεί να σκόσετε το χέρι, μια μικρή προσπάθεια χρειάζεται. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τι να πω για την ομάδα σας κύριε τα τέλος πάντων. Λοιπόν, 57 τροπολογία και υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ, εγκρίνεται. 17 της ηγητή για να βγουν οι λέξεις The Union. Ψήφι υπέρ. Κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αποχές εγκρίνεται. 58 Brandner. Μας λένε εδώ ότι είναι out of budget scope. Τέλος πάντων. Ο συγκεκριτής είναι αντίθετος. Ψήφι υπέρ. 1, 2, 3. Κατά. Πολύ. Αποχές απορρίπτεται. 59 Νιένσκι. Ο συγκεκριτής υπέρ. Ψήφι υπέρ κατά αποχές όπως και πριν. Εγκρίνεται. 18 του ηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. 1, Αποχές εγκρίνεται 20 του εισηγητή με την προφορική τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. 1, 4, 5. Αποχές εγκρίνεται. 61 λοιπόν, η 61 καταπίπτει. 21 τροπολογία του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές είναι κατά. Λοιπόν, τότε να το επαληθεύσουμε. Κάντε προσπάθεια όμως κύριοι συνάδελφοι, να σηκώνετε ψηλά το χέρι να σας βλέπω. Για την 21 ψηφίζουμε τη συγητή ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιοι συνάδελφοι κοιμούνται σήμερα. Να μην πω και ποιοι είναι αυτοί, ε, τέλος πάντων. Λοιπόν, Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν στο τσακ. 62 Μπραντνερ, ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι υπέρ, αλλά θα το ελέγξουμε για μια ακόμη φορά. 62. Σφραντσέσκα. Πέρας ψηφοφορίας. Και όμως, 15 υπέρ, 16 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Α, Ήσασταν υπέρ. Και εσείς. Καλώς. Ας ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, το ακυρώνουμε το αποτέλεσμα και ξαναψηφίζουμε. Για ποια τροπολογία ψηφίζουμε, γιατί το ξέχασα, λέει ο πρόεδρο. Α, την 62, ναι. Γιατί και εγώ τα έχασα. Λοιπόν, 62, 62. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία είναι όμως, άρα απορρίπτεται. τέλο πάντων πάει κάποιες πολιτικές πολύ λεπτές αποχρώσεις εδώ, είναι λίγο πολύπλοκο. Όπως και να έχει, η Φραντσέσκα θα τα βρει εκεί με τους δικού. Λοιπόν, τροπολογία 63, Νιένσκι. Έχει προσερθεί το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64, Νιένσκι. Ο εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 της Φραντσέσκα Μπραντνερ. Ο εισηγητής είναι αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία 66 της Φραντσέσκα Μπραντνερ σε δύο τμήματα, για το οποίο και ο εισηγητής είναι και στα δύο αντίθετος. Πρώτο τμήμα, χωρίς τις λέξεις The Peace Building. Δεν θέλει ειρήνη η Φραντσίσκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Η ειρήνη μπαίνει εδώ, αλλά πάλι δεν τη θέλει. Τέλος πάντων. Ποιοι είναι υπέρ των λέξεων αυτών The Peace Building. Τρεις κυρίες είναι υπέρ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κατά. Πάει. Λοιπόν, τροπολογία και 67 νιέν. και ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 με το δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί. Περ κατά, ε, ένας. Όχι, τέσσερις κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 τροπολογία του εισηγητή. Ψήφι περ. Κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αποχές εγκρίνεται. 69 Νιένσκι συμβατή εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Η Γιούτα είναι κατά, άρα θα πρέπει να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 69. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. 23 του εισηγητή, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 του εισηγητή, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70. 71 μπορούμε να τις πιέσουμε και τις δύο μαζί. Ωραία. Η συγκητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Τέσσερις. Αποχές. Εγκρίνονται και οι δύο τροπολογίες. 25 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 του Σάρλ Γκέρενς. Ο εισηγητής υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε στα παραρτήματα. 73 τροπολογία από την ΚΟΕ. Ο συγγετής αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Περίεργη αυτή η πλειοψηφία. Εγώ λέω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θέλετε να ψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες της ΚΟΕ μαζί. Α, όχι. Όχι, όχι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, ή τουλάχιστον τις έξι πρώτες, δηλαδή 73 έως και 78 που ο εισηγητής είναι αντίθετος. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε από κοινού αυτές. Ηλεκτρονικά, έτσι, για να είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 73, την 74, την 75, την 76, την 77 και την 78 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ 15 κατά. Εγκρίνονται όλες αυτές οι τροπολογίες. Άλντα Ντεσάζα, συγχαρητήρια. Πάμε στην 79, εδώ είναι πιο πολύπλοκο. Έχουμε και ε, τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, από το κομμάτι που λέει Supporting Specific Initiatives μέχρι το κομμάτι National Health Policies που δεν αρέσει τον εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές, ή πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμφιλίωση για το δεύτερο τμήμα. Να ψηφίσουμε τώρα τις τρεις επόμενες 80, 81, 82 μαζί. Διανατάσσος ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς δεν άλλαξε γνώμη έτσι. Θρίαμβος. Θρίαμβος για την ΚΟΕ. Συγχαρητήρια. Πάμε στα recitals, σε αιτολογικές σκέψεις. 3-4-5 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 28-29 Μπραντνερ από κοινού. Όχι, δεν θέλετε. Δεν θέλετε. 28 καταρχάς λοιπόν, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 της Μπραντνερ πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 συμβατή τροπολογία. Εισηγητής είναι αντίθετος όμως. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ θα προτιμούσα, επειδή υπάρχουν πολλοί που απέχουν, να το ελέγξουν ηλεκτρονικά. Τροπολογία 30. Μπραντνερ. Πέρας ψηφοφορίας. 11 υπέρ 17 κατά 5 αποχές απορρίπτεται. 31 Μπραντνερ. Εξωγή είναι και αυτή η τροπολογία. Κατά ο εισηγητής ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 32 Μπραντνερ. Ο εισηγητής αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή τη φορά εγκρίνεται. Ρευστές οι πλειοψηφίες. Λοιπόν, 33 μονήθηκε εξωγήινοι και αυτή. Ο συγητής όμως την υποστηρίζει αυτή την τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ε, ναι. Αποχές εγκρίνεται. 34 του κ. Χάρτονγκ. Ο συγητής είναι αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πιο πολύ. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. 35 Μπραντνερ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Από την ΚΟΕ. Εξωγήινη τροπολογία, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Άλντα, ε, δεν σου μπορεί να το αισθανθεί κανείς σήμερα. 37 Φραντσίσκα Μπραντνερ, ο σχετής αντίθετος, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, κατά, με μικρή διαφορά απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές υπέρ αυτή τη φορά πιο πολύ, άρα εγκρίνεται 39 της Μαρία Μουνίπ συμπατεί με την 38, ο ηθοσυγητής αντίθετος ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 40 Μπραντνερ, ηθοσυγητής αντίθετος ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 Το κύριο Χάρτον, εισηγητής αντίθετος, υπέρ, 3. Κατά, περισσότεροι. Αποχές, απορρίπτεται. Η 42 της κυρίας Μουνίθ, κατά τμήματα, ο εισηγητής είναι υπέρ και των δύο. Πρώτο τμήμα, Fighting Climate Change έως Reinforce Their Impact, ψήφι υπέρ, κατά, 8. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, notwithstanding the fact, μέχρι and additional. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. 43. Out of scope και αυτοτροπολογία της κυρίας Θεώρηση για τις αντίθετος ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 44 του Λούκας Χάρτον, ψήφι υπέρ. 3. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, περνάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 1 και 2 του εισηγητή. Λοιπόν, ωραία. Ψήφι υπέρ. Κατά. 4. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 26, Μουνίθ, συμβατή με την τροπολογία. Δεν είναι υπέρ όμως εισηγητής. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27, Χάγλουντ Γκέρενς. Συμβατή αντίθετος εισηγητής. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται γιατί τα μαμούθ είναι κατά. Κύριε Σιγητέ, θέλετε το λόγο. Μπορούμε να ελέγξουμε, σας παρακαλώ, την τροπολογία 48, αν έχει εγκριθεί, αν έχει απορριφθεί. Την 48 παρακαλώ. Τη 48 λέει ο πρόεδρος. Για να δούμε. Η 48 στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της Μαρία Μουνίθ, μάλιστα. Για να δούμε. Τι λέει η γραμματεία. Η γραμματεία έχει ότι εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε, μήπω. Στην αρχή δεν λέτε για το άρθρο 2 παράγραφος 2. Ο εισηγητής ε, δεν είναι βέβαιος. Εγώ θα έλεγα μπορούμε να ξαναψηφίσουμε, αν συμφωνείτε, την 48 της Μαρία Μουνίθ. Συμφωνείτε? Λοιπόν, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Mm. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 16 κατά. Αποχές κτλ. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε η τροπολογία 48. Καλά κάναμε και το ελέγξαμε γιατί έγιναν και κάποιες αλλαγέ. Τελική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. «28 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στο Γιάνν Κοσλόφσκι». Έγιναν δεκτές δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις του. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, πού περνάμε, στο σημείο 23. Είναι το πίσω του Ταμείου Προσάμιση στην Παγκοσμιοποίηση. για την ε, για, το, για την οντέση της Δανίας, το Όντενσε και θέλει ο εισηγητής να μας πει κάποια πράγματα. Ε, η, το αίτημα αυτό είναι σύμφωνα με τις διατάξεις μας πρόκειται για μεγάλο ναυπηγείο προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας πολλά δεξαμενόπλια και άλλα πλοία τα τελευταία 100 χρόνια κατασκευάστηκαν εκεί Τώρα κατασκευάζονται στην Κορέα και στην Κίνα τα πλοία και το ναυπηγείο έκλεισε πολλοί ε, τεχνίτες, ναυπηγοί και άλλοι σιδηρουργοί έχασαν τη δουλειά τους και τώρα πρέπει να επανακαταρτιστούν για να βρουν ένα νέο μέλλον και νέες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεγητά. Έχουμε αρκετές τροπολογίες. Τροπολογία 2. Καλύπτεται από την πρώτη παράγραφο. Δεν το ψηφίζουμε. Θεωρούμε ότι λαμβάνεται υπόψη. Τροπολογία 3. Που καλύπτεται από την παράγραφο 2 του σχεδίου έκθεσης. Εκτός από το δεύτερο τμήμα καλεί την Κομισιόν urges the, commissions, the Commission μέχρι το occasions για να αντικαταστήσουμε τη δεύτερη φράση της παραγράφου 2. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά. Η πράσινη υπέρ ή κατά. Χέλγκα, τι είσαι, υπέρ ή κατά. Υπέρ. Αποχές. Υιοθετείτε το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 4 των φιλελεύθερων. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία απορρίπτεται. 5 της Περβάνς Μπερές και άλλων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 5, 6, 7 μαζί που είναι των ιδίων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Όχι. Ο Αν Γιάνσεν Όσο λέει όχι, τόσο τη βρίσκει. Υπέρ, η πέντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Η έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Εφτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. είχαν διαφοροποιημένη θέση φιλελεύθερη όμω Σωστό είναι αυτό. 8. Των φιλελεύθερων. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ από εσά. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Η 9. Δεν ψηφίζουμε γιατί καλύπτεται από την παράφο 9. 10. Ο εισηγητή είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Η φιλελεύθερη και η συντηρητική. Άλλος κατά. Όλοι οι υπόλοιποι Απορρίπτεται. Η 11 της Pervenche σε δύο τμήματα. Ο εισηγητής είναι υπέρ της, του πρώτου τμήματος. Ποιος είναι υπέρ από σας. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Το δεύτερο τμήμα. Especially weak. Που δεν του αρέσει το εισηγητή. Δεν του αρέσει η αδυναμία. Υπέρ κατά αποχές παρά τις προσπάθειες του Γκέραν ο Γκέραν έπεισε τους πράσινους αλλά όχι τους αριστερούς απορρίπτεται λοιπόν 12 ο εισηγητής είναι υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές υιοθετείται 13 των φιλελεύθερων ο εισηγητής είναι κατά υπέρ παρακαλώ φιλελεύθερη και συντηρητική κατά οι περισσότεροι απορρίπτεται. 14. Της Περδόνς. Ο εισήτης είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Η ίδια πλειοψηφία πάνω κάτω μου φαίνεται. 15. Της Περδόνς. Ο εισήτης είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 της Περδόνς. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ από εσά κατά, αποχές, υιοθετείτε. 17 των φιλελεύθερων. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Το ΕΛΚ θα πρέπει να είναι υπέρ, δεν, δεν θα έπρεπε. Όχι, καλά. Κατά. Συγγνώμη. Τα μαμούθ κάνουν σκόνη τους φιλελεύθερους. Τελευταία τροπολογία, νούμερο 1, των φιλελεύθερων εισηγητής είναι κατά. Κατά. Τα ίδια απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα 28 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα. Για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Του Ναράγχο Εσκομπάρ. Του δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για ένα λεπτό θέλω να δώσω κάποιες πληροφορίες που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το αίτημα για κινητοποίηση 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αραγωνία στην Ισπανία. Η ανεργία εδώ έχει πολλαπλασιαστεί, έχει τριπλασιαστεί. 15% όλων των ανέργων βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, η οποία επλήγει σκληρά όπως και ε, στον, αυτο... στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το τομέα των ακινήτων και υπάρχουν ανισορροπίες. Ο κατασκευαστικός οικοδομικός τομέας ε, πλήγει σκληρότατα και καταστράφηκαν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, καταβαραθρώθηκε η απασχόληση. Όλος ο οικοδομικός ε, τομέας επλήγει σκληρά και όλοι οι άλλοι τομείς ε, στις 28 Δεκεμβρίου πέρσι αρχίσαμε ένα πακέτο. Οι ισπανικοί οι ισπανικές περιφέρειες προσαρμόζονται ε, με περικοπές για να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα. Μιλάμε για περικοπή στην παραγωνία 500.000 και το εισόδημα έπεσε κάτω από το μέσον όρο στην Ένωση για πρώτη φορά από το 2001. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κινητοποιηθεί το μέσο αυτό. Θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία που περιθωριοποιεί κοινωνικά. Ε, παρακαλώ να το στηρίξετε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Muchas gracias, λέει Πρόεδρος. Οι τροπολογίες 2, 3 και 4 δεν χρειάζεται να ψηφιστούν γιατί καλύπτονται η πρώτη από την πρώτη παράγραφο, τη δεύτερη από τη δεύτερη παράγραφο και η τρίτη από την τέταρτη παράγραφο του σχεδίου έκθεσης. Μιλάμε για τη σχέση μεταξύ της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Επομένως, ψηφίσουμε την πέντε του Αλεξάνδρ Άλβαρο. Η είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 της Περβάνς υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ επίσης. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Η 7. Λαμβάνεται υπόψη από την παράγραφο 5. Δεν ψηφίζουμε. Η 8. Του Άλβαρο. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 9 της Περβάνς που καλύπτεται από την παράγραφο 7 εκτός από το κομμάτι που λέει in order to improve κτλ. Προκειμένου να βελτιώσουμε την ε, σχέση ανάμεσα στην αγορά και στη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 10. Της Περβάνς. Ο εισήτης είναι υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές Υιοθετείτε. Η 11 της Περβάνς με προφορική τροπολογία που αντικαθιστούμε το regrets με το notes. Υπέρ παρακαλώ, κατά, άποχες, υιοθετείτε. Ξεχνάμε τις α, τύψεις. Η 12 του Άλβαρο, ο εισήτης Κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Τα μαμούθ το σκότωσαν το σημείο αυτό. Τροπολογία 13 της Περδόνς, Ο εισήτης είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Υιοθετείτε. 14 της ε, Περδόνς, Ο εισήτης είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια πλειοψηφία υιοθετείται. 15 του Άλβαρο. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ, παρακαλώ από εσά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία 1 του Άλβαρο. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Κύριε Ναράγχο Εσκοβάρ. Και πάμε τώρα στην ψηφοφορία για τις δύο εκθέσεις της Μπάρμπαρα Ματέρα, που είναι πάντα μια στιγμή συγκίνησης. Καταρχάς, η έκθεση κατάρτιση του προγράμματος Δικαιώματα και Ιθαγένεια για την περίοδο 2014-2020. Τροπολογία 25 της κυρίας Βεργιά. Η σχετής είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι η περισσότεροι είναι κατά, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται όντως. Τροπολογία 5. Της εισηγήτριας υπέρ, παρακαλώ, κατά. Αποχές, υιοθετείτε. 26. Βερζιά. Η είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ίδια πλειοψηφία με πριν. 6. τη συγκέντριας. Υπέρ. Κατά. Αποχέ υιοθετείται. Ψηφίζουμε την 27, 28, 29. Δεν θέλετε. 27. κυριε Βεωζία. Η συγκέντρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ κατά εποχές απορρίπτεται 28 ψήφι υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 7 της εισηγήτριας υπέρ παρακαλώ κατά αποχές υιοθετείται 30 Βεργιά. Η συγκέντρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 8. Της συγκίτρια. Υπάρχει ψηφοφορία κατά τμήματα. Αποσύρεται. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα που θέλει να διαγράψουμε τη λέξη corporate. Συμφωνεί η συγκίτρια. Είναι και πρόταση ηγητρίας. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Βγάζουμε τον όρο εταιρικός. Ψηφίσουμε 32, 31 και 32 μαζί. Ναι. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Υιοθετούνται και οι δύο. 33. Γκρέσλε. Υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ από εσά. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 9 της συγκήτριας υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι υπέρ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψηφί υπέρ, 12 κατά. Καμία αποχή. Υιοθετείτε. Η 11. Για τον τίτλο. Βεωζιά. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχή απορρίπτεται. Η 12. Τη κυρίας Βεωζιά. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Η 13. Βεωζιά. Η συγκίτρια κατά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται άνετα. Η 14 βαζία. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές διαθετείτε. 15 βαζιά. Μα είναι αντίθετη γνώμη της συγκήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 16 βαζία, Η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Γκάγκα θα πάλι. να θέμα απορρίπτεται. Ε, αποσύρεται. Ψηφίζουμε όλη την τροπολογία, γιατί δεν προτείνεται η τροπολογία κατά τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες 18, 19, 20 μαζί. Ορισμένοι είναι τόσο κακοί απέναντι στον πρόεδρό του. Έτσι το εξηγώ εγώ. Ψήφιν 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις παρατηρήσεις. 21. Περζιά. Η την είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ από σας. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 3 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Από... Υιοθετείτε. 22 και 23. Να τις ψηφίσουμε μαζί. φυσικά όχι. 22 της κυρίας Βερζιά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές διαλύεται 23 της Βερζιά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά με κομψότητα 4 της εισηγήτριας υπέρ κατά Υιοθετείται 24 της η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Να ψηφίσουμε και τις τρεις μαζί. Α, ναι, ίσως αυτή τη φορά. Α, ναι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετούνται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την πρώτη έκθεση της Μπάρμπαρα Ματέρα. Πέρας ψηφοφορίες, 28 υπέρ, 3 κατά, 2 εποχές. Μπράβο Μπάρμπαρα. Μιλούσαμε για τα δικαιώματα του πολίτη. Χάρη στην Μπάρμπαρα Ματέρα, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν επιτέλους δικαιώματα. Και τώρα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τη δικαιοσύνη για την περίοδο 2014-2020. Άλλη έκθεση της Ματέρα. Τροπολογία 6 της γήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι τροπολογίες ερωτώ της κυρίας Άλντε μπορούν να ψηφιστούν μαζί όλες εκτός της 17. Ωραία, τέλεια. Τι λέτε, τι λέτε να βάλω το 13, τη 14, το 15, όχι, 13 και 14, ωραία. 13 και 14 μαζί, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται οι 13 και 14. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις 15, 16 και 17. 15 και 16, ε, εντάξει. Ψήφι υπέρ, 15 και 16. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της Μπάρμπαρα. Έχει αποσυρθεί, α, όπως και πριν, έχει αποσυρθεί το αίτημα για κατά τη μεταψηφοφορία, άρα ψηφίζουμε απλά για τη διαγραφή της λέξης corporate. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, Απομένως διαγράφει τη λέξη corporate. Τροπολογίες 18-19 μαζί. Ωραία. Ψήφι υπέρ 18 και 19. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 της ηγήτριας, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Αρκετές τροπολογίες πάλι, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Τι κάνουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε από κοινού όλες τις τροπολογίες του Γιούργεν Κλούτε πλην τις 26. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται όλες. Τώρα ψηφίζουμε την 26. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές και αυτή απορρίπτεται αλλά με μικρότερη διαφορά. Ερχόμαστε στις ειδολογικές σκέψεις, τα recital 10 τροπολογία του Γιούργεν Κλούτε είναι υπέρ εισηγητής, αλλά με προφορική τροπολογία, ή εισηγητήρα, συγγνώμη, που μιλά για το Public Awareness Prevention of Drug Trafficking, Illicit Drug Trafficking, Other Illegal Activities Related to Drugs. Ψήφι υπέρ. Κατά. Μόνο η πράσινη κατά αποχές. Ωραία. Άρα εγκρίνεται η τροπολογία 10 με την προφορική τροπολογία. Τροπολογίες 11-12 μαζί μπορούμε. Ωραία. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Τις τροπολογίες της 3, 4, 5 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και εδώ μαζί μπορούμε να ψηφίσουμε τις τρεις τροπολογίες που έχουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Υπέρ, τρεις. Κατά αποχές, ωραία. Εγκρίνονται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε, μην τρέπεστε. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 3 κατά, δύο εποχές συγχαρητήρια στην Μπάρμπαρα. Που έσωσε και τα δικαιώματα των πολιτών και τη δικαιοσύνη ταυτόχρονα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις μεταφορές πιστώσεων. Στις αιτήσει μεταφοράς, λοιπόν. Δεν είναι εδώ η Φραντσέσκα Μπαλτσάνη, αλλά μου έδωσε οδηγίες. Άρα, θα σας ε, μεταφέρω εγώ τις προτάσεις της ε, Φραντσέσκα, εκτός μήπως θέλει κάποιος από την ομάδα της να την αντικαταστήσει. Όχι, άρα εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, σας υποβάλλω τις εξής προτάσεις. Αν τώρα δεν έχω καταλάβει καλά τι μου είπε η Φραντσέσκα, μην διστάσετε να με διορθώσετε. Πρώτον, δύο μεταφορές, 11 και 14, που αντιστοιχούν στις ψηφοφορίες που είχαμε πριν για την κινητοποίηση συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου που προσαρμόζει την παγκοσμιοποίηση. Εγώ λέω να ψηφίσουμε μαζί αυτά τα δύο. Υπέρ των μεταφορών αυτών. Κατά αποχές εγκρίνονται. Και είναι και απόλυτα λογικό. Τώρα, ΔΕΚ 19. Πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ε, γιατί πετύχαμε στη Διελγιστίνα που είχαμε με το Συμβούλιο Πετύχαμε λοιπόν και επικρατήσαμε για το κατά πόσο θα έπρεπε τα 508 περίπου εκατομμύρια ευρώ που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί από τα προηγούμενα έτη για την έρευνα. Ξέρετε ότι αρχικά ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικό το Συμβούλιο και χρειάστηκε να αναφέρουμε το ότι είναι πιθανό το Κοινοβούλιο να μην ψηφίσει τον τελευταίο διορθωτικό προπολογισμό του 2011 για την επιστροφή των πλεονασμάτων του προπολογισμού του 2011 στα κράτη-μέλη. Και έτσι άλλαξε στάση στο Συμβούλιο. Άρα με τη μεταφορά αυτή μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα όπως το επιθυμούσαν. Η εισηγήτρια λοιπόν θερμά μας παροτρύνει να στηρίξουμε αυτή τη μεταφορά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές, επομένως εγκρίνεται. Τώρα μεταφορά DEC 21 για τη χρήση πιστώσεων, για την ανθρωπιστική και πιστιστική βοήθεια της ανάγκης. Δεν φαντάζομαι ότι εδώ έχουμε πρόβλημα. Η συγγήτρια μας ε, συνιστά να ψηφίσουμε υπέρ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, επομένως εγκρίνεται αυτή έτσι μεταφοράς. Υπάρχει επίσης το ΤΕΚ 18. Δεν το έχουμε στον κατάλογο του Κόμπου News, το έχετε όμως λάβει εκ των υστέρων. Ε, πρόκειται για άρση επιφύλαξη στο προπολογισμό επικοινωνίας, το ζήτησε η Επιτροπή Κουλτ ε, Πολιτισμού. Η σύντρα είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές εγκρίνεται. Τέλος προς ενημέρωση. Να σας πω ότι έχετε στο φάκελό σας την προσαρμογή σε πιστός πληρωμών μεταξύ των ε, τεχνικές δηλαδή προσαρμογές μεταξύ των κονδυλίων για την έρευνα διαβάζω το υπολογισμών για ενημέρωσή μας αυτές τις πληροφορίες. Αυτά για τις μεταφορές πιστώσεων. Σας ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε, αφού ολοκληρώσαμε με την Επιτροπή, στα άλλα τμήματα, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουν ζητηθεί εδώ ε, κάποιες ε, μεταφορές πιστώσεων. Θεωρώ ότι είναι ε, δικαιολογημένες, νόμιμες. Άρα θα έλεγα να ψηφίσουμε υπέρ όλων αυτών των αιτήσεων μεταφοράς. Αν θέλετε μπορώ να σας επεξηγήσω συντομία για την κάθε μία περίπτωση τι γίνεται μεταφορά για το δικαστήριο 172.000 ευρώ για διοικητικούς σκοπούς για τις νέες τεχνολογίες για το δικαστήριο για να βελτιώσει το, τα συστήματα διαχείρισης και υπάρχει και μια άλλη αλλαγή Υπάρχουν 2 για το δικαστήριο 20.000 ευρώ και για το κοινοβούλιο ...230.000 ευρώ για το νέο κανονισμό των μελών στα πλαίσια του νέου κανονισμού και ένα ακόμα 33.770 ε, για συντήρηση, δαπάνες συντήρησης και δαπάνες αλλαγών για την Ευρωπαϊκή και ε, ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μετά για την Επιτροπή των Περιφερειών μια άλλη αλλαγή στον προϋπολογισμό, 16.836 ευρώ που θα καλύψουν ανάγκες συντήρησης και μεταφορές, μετακινήσεις επίπλων και μια άλλη για την Επιτροπή Περιφερειών 17.000 ευρώ για τεκμηρίωση και δαπάνες βιβλιοθήκης. Μετά υπάρχει και μια άλλη αλλαγή για την Επιτροπή των Περιφερειών, 77.000 ευρώ για την ΚΡΕΣ, για τον υπηαγωγείο ή τον βρεθονιπιακό σταθμό. Καλό αυτό για το προσωπικό. καλύπτονται από εκεί, το, καλύπτεται από εκεί ο βρεφονιπιακός σταθμός και νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε ε, υπέρ όλων αυτών των ετοιμάτων μεταφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρα, ο εισηγητής είναι υπέρ όλων αυτών των επτά αιτήσεων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δύο. Αποχές, επομένως εγκρίνονται και αυτά. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Πού πάμε τώρα. Πηγαίνουμε στο σημείο 29. Πολιτική ακινήτων. Θα επανέλθουμε το απόγευμα σε άλλα θέματα, αλλά θα παρακαλέσω τη Μόνικα Χολμάγερ να μας πει κατά πόσον θέλει να ψηφίσουμε για το Gender Institute του Βίλνιους. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσουμε αυτό λοιπόν στα γαλλικά. Μόνικα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι για την ισότητα των φίλων που είναι στο Βίλνιο στη Λιθουανία. Υπάρχει ένα ντοσιέ γιατί ε, έπρεπε να, στα πλαίσια της ίδρυσης να μισθωθούν ακίνητα τα οποία ήταν και οικονομικά στη Λιθουανία το Κοινοβούλιο έχει ένα γραφείο ενημέρωσης, μια αντιπροσωπεία οικομισιών και θα συσταγαστούν. Γι' αυτό έγινε έρευνα αγοράς και θα υπάρξουν συνέργειες και κέρδη και θα καλυφθεί το 50, θα χρειαστούμε το 50% του ακινήτου, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή ε, θέση στο κέντρο του Βίλνιους, ε, ανήκει σε μια θηγατρική του ομίλου IKEA, αποτελείται από δύο ενότητες χωριστά, το ένα είναι ξενοδοχείο και το άλλο είναι ένα shopping mall, το οποίο τώρα θα ε, γίνει γραφεία και εκεί θα μισθώσουμε γραφεία ε, με 10, για 10 έτη με οψιόν διακοπής στα 5 χρόνια θα υπάρξει ένα κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης. Εδώ είναι λίγο περιορισμένος ο χώρος. Εγώ συμφωνώ, εγώ είδα την, τον οριζόντιο κανονισμό που προβλέπει κέντρο τεκμηρίωσης. Ακόμα και αν εμείς το βλέπουμε επικριτικά ως Επιτροπή, αυτή είναι απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει ληφθεί και εμείς δεν μπορούμε να άρουμε τον κανονισμό με αυτά που θα πούμε, θα δεχτούμε προηγούμενες, προηγουμένως αποφάσεις και γι' αυτό και οι, οι χώροι που δεν είναι τεράστιοι για ένα κέντρο τεκμηρίωσης θα πρέπει να ε, γίνουν αποδεκτές ούτω ώστε να μπορεί να γίνει κάποιο, κάποιες από τις εργασίες που έχει. Είναι περίπου 2.000 τετραγωνικό μέτρα το εμβαδόν μέχρι το 2013. Θα είναι 64 ε, εργαζόμενοι εκεί. Ε, υπάρχουν κάποιες δαπάνες που πρέπει να ε, καλυφθούν με βάση τον προϋπολογισμό. Το ενίκιο είναι λίγο χαμηλότερο από ό,τι εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, γίνεται παρατήρηση στην ομιλήτρια γιατί μιλάει γρήγορα. λοιπόν, το ενίκιο θα είναι για 10 χρόνια και συνολικά είναι 4,9 εκατομμύρια ευρώ οι δαπάνες. Πιστεύω, επειδή η τάξη μεγέθους στο μελλοντικό προϋπολογισμό και στη ρύθμιση του δεν θα περνάει εδώ και θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και θέλω να ευχαριστήσω την συνεισηγήτρια από τη σοσιαλιστική ομάδα γιατί χθες ε, της έδωσε η γραμματεία τα έγγραφα. Ελπίζω να γίνεται ε, πιο έγκαιρα η παροχή των εγγράφων. Πάντως, ε, καλό είναι ότι μπορούμε να πούμε ναι. Επίσης ήρθα σε επαφή και με τον ασθενή George Lyon και συμφωνεί και εκείνος. Επειδή ήταν λίγος ο χρόνος, δεν μπορούσαμε να έχουμε πλήρεις επαφές μεταξύ μας και να συνεννοηθούμε. Πάντως γενικά είναι καλή η πρόταση και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, περιμένουμε για έξι εβδομάδες. Καλό είναι λοιπόν ε, να ε, προχωρήσουμε για να προχωρήσουν και οι αρμόδιοι ε, πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Συγήτρια. Η γραμματεία έχει διαβιβάσει τα έγγραφα. Ε, τα διαβίβασε όταν τα έλαβε. Τα λάβαμε αργά βέβαια, αλλά και αυτοί τα έλαβαν αργά. Δυστυχώ. Υπάρχει ένα πρακτικό έτσι πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Λοιπόν, άρα λέει η συγκεκριά μα να δώσουμε πράσινο φω. Μα λέει να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμά μα να δώσουμε γνωμοδότηση. Αν συμφωνείτε λοιπόν, δεν θα ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό. Λήξη λοιπόν των ψηφοφοριών και επαναρχόμαστε στην μέση διάταξη. Τι έχουμε προβλέψει στο σημείο 5. Να συζητήσουμε το πολιτισμο πλαίσιο. Να σας πω εγώ λίγα πράγματα εν συντομία. Κατόπιν αιτήματα των δύο γητών για τις δαπάνες, που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν μπορούν να είναι εδώ, ο Ράιμερ Μπέγκε και ο κ. Κάλφιν, Αν οι συνάδελφοι που είναι αρμόδιοι για τους ιδίους πόρου Ντεάν και Γένσεν, θέλουν να συμπληρώσουν κάτι, ευχαρίστω να το πράξουν. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξή. Τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πρώτη φορά κατάφερε να αναφέρει το πρόβλημα του δημοσιονομικού πλαισίου. Επευκαιρία της συνεδρίασης του της 28-29 Ιουνίου, όπως προβλεπόταν. Όπως επίσης μπορούσαμε να υποθέσουμε το 98% της συνεδρίασης αυτής του Συμβουλίου ήταν αφιερωμένο στην χρηματοοικονομική κρίση και το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο αποτέλεσε ένα αντικείμενο μόνο ενός πολύ γρήγορου γύρου τραπέζης. Τα συμπεράσματα που σας ανέφερα και πριν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσαν το χρονοδιάγραμμα με επιθυμητή καταληκτική μερομήνια πολιτικό στόχο το Δεκέμβριο του 2012 και είναι ένα χρονοδιάγραμμα που με βάση αυτό εμείς δουλεύουμε τόσο καιρό, άρα αυτό επιβεβαιώνεται. Επίσης, η Κυπριακή Προεδρία κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει τώρα διαπραγματεύσεις πιο συγκεκριμένες και εντός Συμβουλίου αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας ως βάση το έγγραφο που ε, ονομάζεται διαπραγματευτικό κουτί και το οποίο είχε υποβάλει προηγούμενη Προεδρία, της Δανίας δηλαδή, όχι όμως ως μόνη βάση εργασίας, μία βάση εργασίας τέλος πάντων θα είναι αυτό το έγγραφο. Επίσης, η Κυπριακή Προεδρία από τη δική της πλευρά δημοσίευσε ένα σημείωμα Φαντάζομαι το έχετε λάβει. Άμεσα το έδωσα το, το διανύμα με στους συντονιστές. Εκεί αναφέρεται ε, το πνεύμα που θα διέπει τι εργασίε τη Κυπριακή Προεδρία και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα σημείωμα το οποίο ανταποκρίνεται σε επιθυμίες του Κοινοβουλίου και ως αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου ε, είχαμε επενθυμίσει και με τους εισηγητές μας σε κάθε συνάντηση με τις τρεις προεδρίες. Τι επιθυμούμε. Και συγκεκριμένα ότι επιθυμούμε να ληφθεί υπόψη η συνθήκη της Λισαβόνας και η πολιτική και νομική θα έλεγα αναγκαιότητα της διάκρισης των θεμάτων που άπτονται του δημοσιονομικού πλαισίου η απόφαση πρέπει να γράφεται στο, στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία και στο κανονισμό για το δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά απ' την άλλη έχουμε και τα θέματα που άπτονται της τακτικής, της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας, ίσως και έκτακτης κάποιες φορές, αλλά εκεί έχουμε συναπόφαση. Η Κυπριακή Προεδρία έλαβε το μήνυμα και το δέχτηκε και καλύτερα από ότι η Ιδανική Προεδρία. Το σημειώνει και στο εγγραφό της, το λαμβάνει υπόψη. Προσεχώς θα έχουμε συνάντηση με την Κυπριακή Προεδρία για να δούμε συγκεκριμένα πώς θα μεταφραστεί αυτό στη μεθοδολογία εργασίας. Η καλύτερη λύση που η ομάδα επαφής προεδρεύοντος του Μάρτιν Σούλτς μου έδωσε εντολή να προτείνω στην Κυπριακή Προεδρία θα ήταν να συμφωνήσουμε να έχουμε αυτόν τον επιμερισμό των θεμάτων. Από τη μία πλευρά τι άπτεται της νομοθεσίας και από την άλλη τι άπτεται του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να φροντίσουμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τις εσωτερικές διαπραγματεύσεις και, την άλλη πλευρά, για τις δικές μας διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών προεδριών και της Αντιπροσωπείας Επιτροπής Προϋπολογισμών, εμείς να μιλήσουμε μόνο για όσα άπτονται του δημοσιονομικού πλαισίου και να παραπέμψουμε στους αρμόδιους σχηματισμούς του Συμβουλίου Υπουργών και στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις διαπραγματεύσεις για τις νομικές βάσεις, για τον κανονισμό, τα ταμεία, τη συνοχή, έρευνα, Ευρώπη στον κόσμο και ούτω καθεξής, ώστε μετά να γίνει μία σύνθεση όλων αυτών αφού θα έχει προχωρήσει απαρκώς η διαπραγμάτευση για την νομική βάση. Ξέρετε ότι σε αυτή τη φάση νομοθετικέ βάσει, ε, τι γίνεται, οι συνάδελφοι των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών θα έχουν ω αναφορά τα στοιχεία τη Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Αυτό το συμφωνήσαμε στην ομάδα επαφή. Λοιπόν, επόμενο στάδιο, 24 Ιανουαρίου. Πρώτη συνάντηση της αντιπροσωπείας μας με τις τρεις προεδρίες. με επικεφάλιση πλέον τον Κύπριο Υπουργό. Τον κύριο Αντρέα Μαυρογιάννη, ε, αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα. Ο ίδιο ε, υπουργό θα είναι και ο συνομιλητή μα για το στο μεσονομικό πλαίσιο, αλλά και για το σχέδιο προπολογισμού του 2013. Ο τριμερή διάλογο λοιπόν που θα ξεκινήσει αρχέ εβδομάδα, ε, που ξεκίνησε μάλλον, είχε ω επικεφαλή των Υπουργών Οικονομικών που μα είπε ότι είναι η πρώτη και τελευταία φορά που μα συναντά και ότι την επόμενη φορά θα είναι ο κύριος Μαυρογιάννης. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο θα διευκολύνει και τις σχέσεις μας με την Κυπριακή Προεδρία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Το τελευταίο που θέλω να σημειώσετε και θα δώσω το λόγο μετά στους συζητητές μας για τους ίδιους πόρους είναι ότι για τους ίδιους πόρους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έκανε κανένα λόγο γι' αυτό, αλλά το ΕΚΟΦΗΝ που προηγήθηκε έκανε λόγο για το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και υπήρξε και ένας γύρος τραπέζης όπου κάθε αντιπροσωπεία, κάθε εθνική αντιπροσωπεία εκφράστηκε, είπε την άποψή της, για το ποιε είναι οι πολιτικέ τη προθέσει, σε ό,τι αφορά την ίδια την αρχή επιβόλη ενό φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Κάποιε αντιπροσωπείε ανέφεραν ότι απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια ιδέα, άλλε αντιθέτω είπαν ότι προτίθενται να εφαρμόσουν αυτή την ιδέα και από εκεί και πέρα Πρέπει να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά το σκέλος ήδη υπόρρη. Τώρα, να δώσω το λόγο στον Ζαν Λουκ Ντεάν, που θα μας παρουσιάσει το πώς έχει κατάσταση και στην Αν μετά. Έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Το μόνο νέο πράγμα για τους ίδιους πόρους χωρίς να ξεχνάμε ότι σε επίπεδο Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων δεν το συζητήσαμε πολύ μέχρι στιγμής, αλλά πετύχαμε από την Ανέσκη Προεδρία στο να μείνει αυτή η σχέση στο διαπραγματευτικό κουτί. Διαπιστώσαμε λοιπόν στο τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ότι δεν υπήρχε πλειοψηφία, εν δεν υπήρχε συνένεση για να βάλουμε το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι αυτό το στοιχείο βγαίνει από τους πιθανούς ιδίους πόρους. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση έχει περισσότερες αποχρώσεις. Και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι είπε ότι η συζήτηση για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν έχει τελειώσει. Και δεν έχει τελειώσει και η συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Θα δούμε τώρα αν η Κομισιόν θα πάρει την πρωτοβουλία για την ενισχυμένη συνεργασία. Και αν θα υπάρξει και μια πρόταση για να διατηρήσει το φόρο αυτό ως τμήμα των ιδιών πόρων, έστω και εν μέρη. Λαμβάνοντας υπόψη την δική μας ε, κατάσταση των συζητήσεων για τους ιδίους πόρους, μπορούμε να διαρωτηθούμε ποια θα είναι η θέση της Κομισιόν επί του φόρου. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι να πούμε ότι όταν θα επεξεργαστούμε το ψήφισμα του Οκτωβρίου, το ενδιάμεσο ψήφισμα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παρότι η νομική θέση σε σχέση με τους πόρους, η θέση μας είναι λίγο διαφορετική, θα πρέπει να κρατήσουμε τη σχέση ανάμεσα στους ίδιους πόρους και στο πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο και σε αυτό το ενδιάμεσο ψήφισμα. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά που θα την κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ, Ζαν αν θες να προσθέσεις κάτι. Uh, Συμφωνώ απόλυτα με τον Ζαν Λουκ. Πρέπει να περιμένουμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και πώς κρίνουν αυτή την κατάσταση όπου κάποια κράτη μπορεί να κάνουν ένα βήμα προς τα μπρος και πώς μπορεί αυτό να καλύψει και την πρόταση για τα, τους ιδίους σπόρους. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε και με την πρόταση για τον ΦΠΑ που δεν ζητεί αλλαγή νομοθεσίας αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή και θα έχουμε πιο πολλές εξουσίες στα εκτελεστικά μέτρα από ότι έχουμε στην πρόταση για φορολογικά θέματα που έχουμε τη διαδικασία των ακροάσεων. Μπορούμε να κάνουμε ίσως κάτι εδώ λοιπόν. Η πρόταση για τον ΦΠΑ όμως είναι αρκετά περίπλοκη, πολύ περίπλοκη, γιατί το σκέλος των δαπανών θα έλεγα ότι ο Ράιμερ και ο Ήβαλο, ο ο Ράι Μπέγκε και ο Ιβαλο Λοκάλφιν είχαν συναντήσει σε μηνιές με τους εισηγητές από τις ειδικέ επιτροπές και έτσι υπάρχει μια καλή εποπτεία των τεκτενομένων στις ειδικέ επιτροπές. Ξέρουμε δηλαδή προς τα πού το πάνε και ε, καθησυχάζουμε βλέποντας ε, την πορεία των εργασιών σε σχέση με τη δική μας προοπτική χρειάζεται πάρα πολύ να έχουμε τη διαδικασία της συναπόφασης και να προχωρήσουμε έτσι και να μην μας ξεπεράσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ξαφνικά από τα πάνω θα υπαγορεύσει μια απόφαση και εμείς δεν θα έχουμε δυνατότητα και εξουσίες. Από την άλλη ακούω και στη δικιά μου την ομάδα κάποιες ανησυχίες τώρα ότι όλα θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα και να τελειώνουν με συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης. Αλλά εδώ συζητάμε για την κοινή αγροτική πολιτική την επόμενη 7 ετία. Συζητάμε τα διαρθρωτικά ταμεία για τα επόμενα 7 χρόνια. Είναι τεράστια τα πακέτα αυτά και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά θα γίνουν με τρόπο διαφανή. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εδώ στην προσπάθεια εφαρμογής των και ε, άσκησης των νέων εξουσιών από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και μου φαίνεται ότι δεν βοήθησε πολύ και δεν ήταν καλό συμπαραστάτη στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Πιθανό. Γκέραν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω και να επεκταθώ λίγο σε κάποια θέματα που αφορούν τη διαδικασία από εδώ και πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να προχωρήσει η διαδικασία, να γίνουν κάποια πράγματα, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με το χρόνο. Είδα το έγγραφο που αναφέρατε ε, της Κυπριακής Προεδρίας για την οργάνωση των εργασιών για το δεύτερο εξάμεινο του 2012 και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα εδώ που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Προτείνουν πρώτον οι συζητήσεις στα άλλα συμβούλια, εκτός από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, να μην οδηγήσουν σε συμπεράσματα ε, ή να προδικάσουν το αποτέλεσμα της οριζόντιας συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι αντιφάσκη εν μέρη σε αυτό που αναφέρω στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τονίζουν την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις συναπόφασης πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να επιτυγχάνουμε κάποια συμπεράσματα, όχι στα ανώτατα όρια, στο πολιετές, αλλά σε όλα τα άλλα θέματα πρέπει να μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Λένε επίσης και δεν μπορούμε νομίζω να το δεχτούμε ότι θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε ε, ακροάσεις στην αρχή μετά με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων κάθε φορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην περιοριστούμε σε ενημερώσεις πριν και μετά, αλλά να μιλήσουμε για διαπραγματεύσεις. Η προετοιμασία για διαπραγματεύσεις πρέπει να πάμε μπροστά όχι να μας ενημερώνει μία πλευρά, να μας ενημερώνει το Συμβούλιο, εμάς το Κοινοβούλιο. Τέλος, λένε στο έγγραφο αυτό ότι η Προεδρία θα συνεχίσει εντατικές εργασίες επί των προτάσεων στοχεύοντας σε μια μερική γενική, μερικός γενική, partial general λέει, τι σημαίνει αυτό Parcel General, νομίζω ότι είναι αντιφατικέ οι έννοιε, τέλο πάντων. Και ταυτόχρονα να κάνει άτυπο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλε τι τομιακέ νομοθετικέ προτάσει. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα άτυπου διαλόγου. Αυτά είναι θέματα χαρτο... συναπόφασης. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι είναι σημαντικό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, όχι ομιλίες και διάλογος και ενημέρωση τώρα θα πρέπει να κάνουμε πραγματικές γνήσιες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ Γκέραν. Αυτά θα πω και εγώ στην Κυπριακή Προεδρία. Ιζαμπέλ Ντιουχόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό σε ένα τόσο λεπτό και δύσκολο θέμα όπως είναι οι ίδιοι και οι σχέσεις τους με το πολιετές να πούμε ότι ε, εγώ συμφωνώ με τον Ζαν Λικ Ντεάν, με τον Γιάν Χάνσεν και με άλλους. Πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε τη σχέση, ώστε να τον πιο πολύ και ώστε να τον πιο για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο φόρο και στο πολιετές. Παρότι ξέρουμε αυτά που ξέρουμε το Συμβούλιο, παρότι περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν για μια ενδεχόμενη ενισχυμένη συνεργασία. Εν συνεχεία θα θα περπατήσουμε πάνω σε μια λεπτή γραμμή για να κρατήσουμε τις διαδικασίες μας, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε εκεί που έχουμε δύναμη. Για την διάμεση έκθεση για το πολιετές πλαίσιο, εκεί είναι πράγματα που έχουμε να πούμε πράγματα. Εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε. Ε, όλα τα υπόλοιπα είναι προφορικές δηλώσεις, περιορισμένης εμβέλειας. Ελπίζω ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι Δηλαδή θα ακολουθήσουμε την Κομισιόν, θα την υποστηρίξουμε στην πρότασή της να κρατήσει οπωσδήποτε την αρχή των ίδιων πόρων που συνδέονται με το πολιτέ πλαίσιο. Αυτό είναι εκ των ονουκάνευ. Παρότι θα πρέπει ήδη μετά τις διακοπές να παρακολουθούμε την εξέλιξη εβδομάδα με εβδομάδα και να δούμε τι θα προκύψει, τι νέο θα έχουμε και από την ομάδα επαφή μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ. Σαλβατόρ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω μόνο γιατί με τις σκέψεις των συναδέλφων συμφωνώ. Τι ενδιαφέρει και τι ε, σχεδιάζει, τι ενδιαφέρει την Κυπριακή Προεδρία και τι σχεδιάζει, αυτό είναι το ερώτημά μου. Είδαμε με τα διαπραγματευτικά κουτιά, με τις διαδικασίες ε, στην απόφαση με το Κοινοβούλιο, φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο το σχέδιό τους. Εκεί θέλουν να συνεργαστούν, σαφώς. Ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, Διαφάζοντα ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης, τι παραπάνω μπορούμε να ελπίζουμε από τις 6 μήνες της Κυπριακής Προεδρίας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει πραγματικά πρόοδος ή αυτό το οποίο περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η τελεία και η παύλα του σχεδίου εργασίας ε, της Κυπριακής Προεδρίας. Δεν θα υπάρξει τίποτε άλλο. Θα υπάρξουν κάποιες ε, διαβουλεύσει μεταξύ των διαφορών αντιπροσωπιών στο Συμβούλιο. Κάποια διαβήματα ίσως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατυπώσει προτάσεις. Ή απλά θα μείνουμε σε αυτό το αίτημα για πιθανή ενισχυμένη συνεργασία. Δεν ξέρω. Να μας πείτε τι βλέπετε. Για αυτό το σημείο, Σαλβαντόρ. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα θα τα θέσω και εγώ στην Κυπριακή Προεδρία για την ε, υπόθεση των ιδίων πόρων είμαστε σε περίεργη κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μίλησε για αυτό το θέμα. Το ΕΚΟΦΗΝ μίλησε. Έξι μισή τουζίνα αντιπροσωπείες ή λίγο παραπάνω είπαν ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στη δημιουργία ενό φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Είναι το μόνο σημείο των ιδίων πόρων για το οποίο μίλησα μέχρι στιγμής αλλά κάτι πολύ πιο αναπάντεχο και που είναι θετικό σε σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι εννιά αντιπροσωπείες που ενδεχομένως ακολουθούνται και από άλλες ή θα ακολουθηθούν σε λίγο χρόνο είπαν ότι από πλευράς τους ό,τι και αν συμβεί θα εφαρμόσουν, θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έτσι λοιπόν ξαφνικά η Επιτροπή αντέδρασε αμέσω και είπε ότι αν ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δημιουργηθεί στα πλαίσια μιας ενισχυμένης συνεργασίας, δηλαδή η διαδικασία προβλέπει συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τα έσοδα από αυτό το φόρο, τουλάχιστον εν μέρη, να θεωρηθούν ως νέος ίδιος πόρος. Αυτή η κατάσταση τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί πολιτικά. Δεύτερον, θα πρέπει να μελετηθεί νομικά. Μπορούμε να κάνουμε την ισχυμένη συνεργασία και να δημιουργηθεί αυτός ο ίδιος πόρος. Και αν ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένας πόρος που σημαίνει νέος φόρος ε, για μια χώρα στα πλαίσια μιας ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά που δεν εισπράτεται ως ευρωπαϊκός φόρος και στους 27, αν θα μπορεί να είναι ίδιος φόρος. Ε, θα πρέπει λοιπόν και νομικά και πολιτικά να το διευκρινίσουμε. Από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί η συζήτηση. Και μέχρι στιγμής το πράγμα έχει προχωρήσει πιο θετικά από το ζήτημα των δαπανών. Ούτως ή άλλως το ερώτημα αυτό θα το θέσουμε στην Κυπριακή Προεδρία και στην Κομισιόν. Εξάλλου, όπως είπαν οι συγητές και όπως είπε και η Ιζαμπέλ για τους νέους ιδίους πόρους, δεν προβλέπεται μόνο φόρο από το χρηματοπιστωτικό συναλλαγών. Ε, η Κομισιόν μίλησε για το ΦΠΑ και είπαμε ότι αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με βάση αυτές τις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τις ξαναζητήσουμε να κάνει νέες που θα δικαταστήσουν τις παλιές αν δεν περάσουν οι παλιές. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτή τη γραμμή και ως προς το χρονοδιάγραμμα παραμένουμε στη βασική θέση του Κοινοβουλίου ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να συμφωνήσουμε τον επόμενο Δεκέμβριο, αλλά αν δεν υπάρξει συμφωνία για τους ίδιους πόρους, θα υπάρξει συμφωνία για τις δαπάνες. Κάτι που με διασκεδάζει εκ των προτέρων είναι αυτό που θα συμβεί, τι θα συμβεί μάλλον, όταν το θέμα των πόρων θα συζητηθεί στο Συμβούλιο. Σε υψηλότερο επίπεδο, στη Σύνοδο Κορυφή δηλαδή. Γιατί όσοι είμαστε σε επίπεδο υπουργών προπολογισμού, οι υπουργοί προπολογισμού θα παντού, εκτός από ορισμένε χώρες, για λόγους πολιτικής αρχής. Αλλά στις χώρες που είναι υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου φόρου επιτοχρηματοπιστωτικών συναλλαγών, οι υπουργοί αυτοί οικονομικών έχουν σαν στόχο πρώτον να παγώσουν ή και να μειώσουν τη συνεισφορά των εθνικών τους προϋπολογισμών στην χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και να πάρουν το σύνολο των πόρων από το νέο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για να χρηματοδοτήσουν ειδικότερα και αποκλειστικότερα τα εθνικά τους σχέδια και τις, ειδικε... και τις ε, εθνικές τους ανάγκες. Και σε πολλές χώρες οι ανάγκες αυτές είναι πολλές και δύσκολες. Ελπίζουν λοιπόν. Υπάρχει μια φόρμουλα στη Γαλλία μάλιστα. Όταν κάποιος ελπίζει να κερδίσει πολλά και από παντού, λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε και την πίλτα ολάκερη που φτιάξαμε και το σκύλο χορτάτο που ταΐσαμε. Πρέπει να διαλέξουμε. Θα πρέπει να διαλέξουν και οι Υπουργοί Οικονομικών. Εάν αυτό που θα κρατήσουμε, που θα διαλέξουμε, θα είναι αυτό που είπε το Κοινοβούλιο από την πρώτη μέρα και αυτό που υπενθυμίζουμε σε όλες μας παρεμβάσεις. Επίσημες και άτυπες, δημόσιες, ιδιωτικές, γραπτές, προφορικές. Οι νέοι διπόροι θα πρέπει να συνεισφέρουν στη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών. Αυτή, σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη-μέλη έχουν την εγγύηση ότι οι ίδιοι πόροι θα εξυπηρετήσουν τους εθνικούς προπολογισμού, θα τους απαλλάξουν από την συνεισφορά τους στις ευρωπαϊκές πολιτικές, από τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αλλά δεν μπορούν να κερδίσουν δύο φορές οι Υπουργοί Οικονομικών. Μπορούν να κερδίσουν μία φορά. Είναι ένα επιχείρημα που δεν μπορεί να καταλάβει ένας υπουργό Οικονομικών. Είναι γενετικό το πρόβλημά του. Ειδικά οι υπάλληλοι έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα γενετικά. Δηλαδή, οι υπάλληλοι των Υπουργείων Οικονομικών έχουν αυτό το γενετικό πρόβλημα. Και έπαθα ε, μετάλλαξη όταν ήρθα εδώ. Ε, οι Πρωθυπουργοί όμω έπαθαν τη μετάλλαξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλόπνου στόχους για την ε, στήριξη τη ανάπτυξη, την ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση το πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε οικονομίες επί των εθνικών προϋπολογισμών, δηλαδή περικοπές, είναι προφανές ότι ο μόνος τρόπος για να τετραγωνίσουμε τον κύκλο είναι να δημιουργήσουμε νέους πόρους που θα τροφοδοτήσουν απευθείας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις ευρωπαϊκές πολιτικές που θα αφορούν ε, μάζες του ευρωπαϊκού πληθυσμού για να έχουμε την απαραίτητη κρίσιμη μάζα ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικές. Και θα απαλλάξουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς από τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών. Μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αλλά μπορούμε να πούμε ο τρόπος με τον οποίο η Δανέζικη Προεδρία, παρά την εχθρότητα της α, κυβέρνησής της για την ιδέα του φόρου, κατάφερε να κάνει την ομάδα να δουλέψει επί του φόρου μας επέτρεψε να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε για αυτό το κομμάτι της διαπραγμάτευσης που είναι πολύ δύσκολο και που στο τέλος, όπως ξέρουμε, θα είναι τελικά το πιο δύσκολο. Ας κρατήσουμε όλα αυτά για αυτό το σημείο της διαπραγμάτευσης, για το δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί έχουμε και πολλά άλλα θέματα στη μέση και θα το συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα και στους συντονιστές, αλλά και στην Ολομέλεια και στην, Επιτροπή, στην Ολομέλεια μάλλον της Επιτροπής Προπολογισμών από το Σεπτέμβριο και μετά, όταν ξεκαθαριστούν τα πράγματα για το πώς θα πορευτούν με την Κυπριακή Προεδρία και όταν θα έχουμε και από το Συμβούλιο κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα. προτείνω τώρα να περάσουμε στις τρεις, εκθέσεις που είχαν προετοιμαστεί από τον Καρλ Χέγκλουντ Χάγκλουν και που τις ανέλαβε ο διάδοχος του κ. Στόρβαλτ για την έρευνα. Παρουσιάστε και τις τρεις εκθέσεις μαζί. To, Να έχουμε μια κοινή συζήτηση και για τις τρεις εκθέσεις που συνδέονται η μία με την άλλη ούτως ή άλλως. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που συνεχίζω τη δουλειά που άρχισε ο, προ... προκάτοχός μου. Δεν θα επιδείξω την ίδια γοητεία ε, όπως ε, εδώ, σε αυτή τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, αλλά όπως είπε και ο Πρόεδρος, τα θέματα είναι αλληλένδετα. Πολύ σε μεγάλο βαθμό συνειφασμένα τα τρία αυτά θέματα. Γι' αυτό θα τα παρουσιάσω από κοινού. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την εξαιρετική πρόταση την Κομισιόν που αντικατοπτρίζει και αυτά που έλεγε από πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αύξηση χρηματοδότησης, ε, απλούστευση κανόνων, ε, μείωση του κενού μεταξύ έρευνας και ενοτομίας, αύξηση των επενδύσεων για να έχουμε συνέργειες στον τομέα αυτών. Σε ό,τι αφορά το Horizon 2020 έχω τρεις βασικές προτάσεις. Θέλω να δούμε τον εγγενή κίνδυνο του συνδυασμού συνοχής και αριστείας στις δύο φιλοσοφίες που είναι σημαντικές. Η αριστεία πάντα πρέπει να είναι η διέπουσα αρχή. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και θέματα ταξινόμησης ή κατάταξης της αριστείας γιατί από ό,τι ακούω από τα πανεπιστήμια όλα παίρνουν ε, τα δέκα σημεία και μετά είναι δύσκολο να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος από τους άλλους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο σαφείς. Δεύτερον, για να εγγυηθούμε στις χώρες, ότι οι χώρες που δεν είναι στη συνοχή δεν θα εξαιρούνται από όλες τις μορφές υποστήριξης ε, της έρευνας, θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, την εμβέλεια των υπαρχόντων μέσων για να συμπεριλάβουμε ένα μεγάλο φάκελο έρευνας ε, ε, και ε, ε, ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων υποδομής. Το EIT πρέπει να έχει πλήρη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της και όχι μόνο τη μισή που η πρόταση είναι να πάρουν τα μισά χρήματα στην αρχή και μετά ανάλογα με την πρόοδο. Αυτό δεν είναι καλό γιατί είναι σαν να δείχνουμε ότι δεν τους εμπιστευόμαστε καθόλου. Να τους δώσουμε όλο το ποσό και μετά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εκτός αυτού υπογραμμίζω τη σημασία της απλούστευσης, του περιορισμού του διοικητικού κόστους, της ενίσχυσης της θέσης των ΜΜΕ και ανάδειξη του κινδύνου στρέβλωσης της αγοράς. Κανόνες συμμετοχής τώρα. Και πάλι η αριστεία υπογραμμίζεται ως η κατευθυντήρια αρχή στις, κατευθυντή... 1 και 13. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τους κανόνες χρηματοδότησης συγκεκριμένα. Ε, προγράμματα κοντά στην αγορά είναι πολύ σημαντικά για τη βασική έρευνα. Ξέρετε τις τροπολογίες όμως εδώ. Απλούστευση των χρηματοδοτικών διαδικασιών, πολύ σημαντικό πράγμα συνήθως ε, υπόκειται σε πρέπει να υπόκειται σε σωστή φορολόγηση. Επίσης ε, στις 4-8 τροπολογίες αναφέρονται θέματα πλούστευσης όπως και στην 9 και 10. Θα πρέπει να υπάρξει το πολιετές αλλά να περιχαρακώσουμε το θέμα της υπέρβασης, να μην υπάρχει υπερβολική υπέρβαση πόρων. Επίσης, ε, νέας γενιάς αντιδραστήρες. Αυτό είναι αντιαμφιλεγόμενο θέμα. Πολλοί θα διαφωνήσουν οι Γερμανοί θέλουν να σταματήσει η χρήση πυρηνικής ενέργειας, πολλοί Γερμανοί. Η προθεσμία κατάθεση των οροπολογίων είναι η επόμενη Δευτέρα. Θα περιμένω τα σχόλιά σας. Και... Μπορεί να χρειαστώ ε, εγώ και οι συνεργάτες μου πιο πολύ χρόνο. Ε, όλες οι ελλείψεις δεν οφείλονται στον προκάτοχό μου, αλλά σε μένα. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ ε, μαθαίνοντας. Είστε πολύ ταπεινόφρονα, αγαπητέ συνάδελφοι. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας και η δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και πολύ σωστά κάνετε και επιμένετε στην ανάγκη να είναι πιο απλή η διαδικασία, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δούμε και αν θα καταλήξει σε μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού μετά από μακρέ διαπραγματεύσει. Συμφώνησαν πλέον τα τρία όργανα. Η συνάδελφο Ινκε ε, Γκρέσλε κάνει καταπληκτική δουλειά και όχι μόνο βέβαια, ε, αλλά ιδίω ε, η συνάδελφο αυτή. Και βέβαια αυτό πρέπει να συμπληρωθεί. Πρέπει να συμπληρωθεί και, για τα, και με τα άλλα προγράμματα. Γκόραν Φέρν. Κάποια αιτήματα Ευχαριστώ για την πολύ καλή παρουσίαση. Ε, μία ερώτηση εσάς και στη Γραμματεία, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν προβλήματα με την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Το νέο μέλος, ε, επίσης, ε, ε, τώρα ανέλαβε το φάκελο. Υπάρχει περίπτωση να παρατείνουμε τουλάχιστον μέχρι Τρίτη το απόγευμα αντί για τη Δευτέρα την προθεσμία κατάθεση. Αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Για κοιτάξτε το. Τώρα, επί της ουσίας, ε, κάποιες παρατηρήσεις και για, ε, απευθύνομαι στη γραμματεία κυρίως ε, και στον εισηγητή. Συγκεκριμένη νομική βάση για το ίτερ. Δεν υπάρχει όμως το πακέτο. Αυτό πώς θα το διευθετήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να γνωμοδοτήσει και για τη νομική βάση του ίτερ η Επιτροπή Προϋπολογισμών. να μας πείτε που, πώς έχει αυτό το θέμα, είναι σημαντικό. Επίσης έχουμε κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την τροπολογία 16 στην έκθεση, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε το θέμα ίτερ. Και υπάρχουν και κάποιες αιτιολογικές σκέψεις, οι 6 και οι 7, στην ε, έκθεση Euratom, που μιλάμε με κάποιο περίεργο τρόπο για το ίτερ. Έχουμε κάποια ερωτηματικά. Λοιπόν, το ίτερ να το κοιτάξουμε λίγο περισσότερο. Κάποια, κάποιες παρατηρήσεις εξ ονόματος ε, της κυρίας Έντιτ Herzog που είναι σκιώδης και μελετά την πυρηνική ασφάλεια στον πραγματικό κόσμο γιατί πήγε στην Ιγναλίνα, είναι στην Ιγναλίνα τώρα στη Λιθουανία με μια αντιπροσωπεία, δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά μου είπε ότι προτίθεται να καταθέσει αρκετές τροπολογίες. Κάποιες έχουν άμεση σχέση με τη βασική προτεραιότητα του εισηγητή το θέμα της αριστείας. Γιατί εκτός από την αριστεία, βέβαια συμφωνούμε απόλυτα ότι η ευρωπαϊκή έρευνα πρέπει να, είναι, να χρειάζεται την αριστεία. Πρέπει όμως να φτιάξουμε και κάποια σύνδεση μεταξύ ε, αριστείας και συνοχής να έχουμε τις, ε, τα σκαλοπάτια για την αριστεία, για ε, περιφέρειες της Ευρώπης που δεν έχουν τις Οξφόρδες και τις Ορβόνες, αλλά θέλουν να τις φτιάξουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, για να έχουμε στρατηγική και γι' αυτό στο μέλλον. Οπότε προτίθεται να καταθέσει κάποιες τροπολογίες εδώ και για την αριστεία, όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και στην καινοτομία και θέλει πολύ να, γίνει μια συζήτηση για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στις εκθέσεις αυτές και θα υποβάλει και εδώ τροπολογίες. Αρχικά το θέμα της συνοχής και η σχέση τη σύνδεση με την ε, αριστεία και την οικοδόμησή της στο μέλλον για μειονεκτικές περιοχές της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Βεβαίω θα ζητήσει σημαντική αύξηση για όλο τον τομέα της έρευνας στα πλαίσια του εβδόμου ου προγράμματος πλαίσιο. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει όταν μιλάμε για απλοποίηση θα υποβάλει ειδικέ τροπολογίες για να δούμε τις δαπάνες του προσωπικού και του, του προσωπικού ε, γιατί και εδώ μπορεί να γίνει απλοποίηση. Προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες για τον κίνδυνο της αφέμαξης εγκεφάλων, brain drain, γιατί υπάρχουν ε, διαφορετικές συνθήκες στα διάφορα, στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Θέλει να μιλήσει για μια ενιαία έρευνα ερευνητών και ερευνών που θα εξασφαλίσει ότι δεν θα φύγουν οι ερευνητέ από τις φτωχές χώρες και θα πάνε στις πλούσιες. Να έχουμε αντί για αφέμαξη κυκλοφορία εγκεφάλων, brain circulation αντί brain drain. Αυτό το θεωρεί πολύ σημαντικό. Θα υποβάλει επίσης και άλλες τροπολογίες για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλπ. Ε, θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες από την ομάδα μας και από την Edith Herzog και ήθελα να παρουσιάσω εξ ονόματός της κάποιες από τις βασικές ιδέες. Σας ευχαριστώ Γκέραν. Θέσατε κάποια ερωτήματα στην αρχή της παρέμβασής σας. Να σας απαντήσω. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, θα μπορούσαμε να την παρατείνουμε για μία μέρα, δηλαδή 17 Ιουλίου αντί για 16 στις 12 το μεσημέρι. Πιο πολύ δεν μπορούμε. Γιατί δεν θα υπάρχει προσωπικό. Αλλά μπορούμε να κερδίσουμε 24 ώρες. Και τα κείμενα, ε, τα έχετε λάβει εδώ και κάποιο καιρό. Φυσικά και θα επαληθεύσουμε το πρόβλημα με τη, βάση, τη νομική βάση για το ΙΤΕΡ. Αν υπάρχει μια συγκεκριμένη επικαιροποιημένη νομική βάση, φυσικά και θα πρέπει να νομοδοτήσουμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπως άλλωστε πράττουμε για τις άλλες νομικές βάσεις. Η Μόνικα Χολμάγερ ζήτησε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, καταρχήν αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Τόρβαλντ δεν τον ζηλεύω. χιλιάδες σελίδες νέων κανονισμών μέσα σε λίγες μέρες που θα πρέπει να κρίνει και να μελετήσει κανείς. Αυτό με ξεπερνάει. Πολύ, πολύ περίπλοκο. Συγχαρητήρια που τα καταφέρατε. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Τέσσερις προ... προτάσεις της Κομισιόν ε, για τα προγράμματα, για τον ορίζοντα 2020, το, την, ε, το Euratom ε, τώρα για την αριστεία και την αρχή της αριστείας πράγματι συμφωνώ πρέπει να την τηρήσω, με έχει δίκιο ο και οι χώρες που δεν είναι τις μη, οι χώρες της μη συνοχής και η διαφοροποίηση για το EIT δεν θα πρέπει να γίνει σε δύο δόσεις η χρηματοδότηση όπως προβλέπει η Κομισιόν αλλά από ό,τι θυμάμαι και από τη συζήτηση, η χρηματοδότηση του EIT από την αρχή θα πρέπει να προβλεφθεί και άλλωστε είναι σημαντικό από την αρχή να προβλεφθούν και να πραγματοποιηθούν αρκετά βήματα. Και εγώ θα κάνω σχετικές προτάσεις. Ε, πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε από, ως Επιτροπή Προϋπολογισμών γιατί δεν θα κάνουμε τη συζήτηση που θα κάνει η Επιτροπή Ήτρε, δεν είναι δυνατόν άλλωστε κάτι τέτοιο. Πάντως αυτό που για μας πρέπει να είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από τα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουμε. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε απλώς εθνικούς πόρους, θέλουμε ευρύτερη προστιθέμενη αξία. Και η αρχή της αριστείας πολύ σημαντικό, δεύτερο είναι αυτό, τρίτον ε, μια διαπαραταξια, ένα διαπαραταξιακό αίτημα είναι η βελτιωμένη πρόσβαση από τις ΜΜΕ στα προγράμματα αυτά, γιατί αυτό εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πάνε κοντά σε μια μεγάλη επιχείρηση να συνεργαστούν, δεν έχουν σχεδόν καμιά ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα. Και κάτι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό για μένα, ε, στις επιδοτήσεις να υπάρχει νομική ασφάλεια και σαφήνεια ε, και στους λογαριασμούς και σε όλα. Γιατί αν έρθουν οι κατευθυντικές γραμμές δύο χρόνια αργότερα και διαφοροποιούνται από αυτά που είχαμε πει στην αρχή και στο τέλος ε, φτάσουμε στα δικαστήρια γιατί δεν θα έχουμε συνεννοηθεί γιατί χρηματοδοτείται κάτι και πώς, αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να το αποφύγουμε. Να υπάρχει νομική ασφάλεια από την αρχή και να είναι ξεκάθαρο ευθύ εξ αρχή τι θα χρηματοδοτηθεί και τι όχι. Γιατί εν μέρη και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα πάμε στα δικαστήρια. Για το ΙΤΕΡ και μένα με ενδιαφέρει να υπάρξει μια διαφοροποίηση του προγράμματος έρευνας και της γραμμής προϋπολογισμού για το ΙΤΑΡ για να μην κάνουμε κάθε φορά τη συζήτηση στο ορίζον 2020 που θα βρούμε τα λεφτά για το ΙΤΑΡ και να τα πάρουμε από εκεί. Πρέπει να έχει αυτόνομη χρηματοδότηση το ΙΤΑΡ, το ερευνητικό του πρόγραμμα. Επίσης, με τα χρήματα που θα ε, ε, ε, πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή επιχείρηση και παραγωγή ε, για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις ε, αποδοτικές μέσα στην Ευρώπη. Τέλος, μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου. Με τη σαφήνεια των κανόνων θα το φροντίσουμε και αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε τεράστιες ε, γραφειοκρατικές δαπάνες και οι ΜΜΕ να μην μπορούν να ε, συμμετέχουν γιατί δεν μπορούν να καταβάλουν τις δαπάνες που είναι συνδυασμένες με μια, ένα τέτοιο πρόγραμμα και τέτοια προώθηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μόνικα Ιζαμπέλ Ντυρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, όπως και άλλοι προλαλήσαντε, στηρίζουμε την πρόταση για σημαντική αύξηση των προγραμμάτων αυτών της κατηγορίας 1α σημαντική προστιθέμενη αξία. Φυσικά δεν θα σας εκπλήξει το ότι θα ζητήσω ε, στεγανή, ε, στεγανή διαχωρισμό ε, για το ίτερ. Διαφωνούμε για το Ευρατόμ, αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμφωνήσουμε ότι πράγματι είναι επίγον και στα ίδια τα προγράμματα να συμμετέχουν οι ΜΜΕ αλλά και στη στήριξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας της ΜΜΕ. Θα κάνουμε επίσης τροπολογίες και σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των σχεδίων. Είναι σημαντικά τα ποσά. Η επιλογή των θεμάτων εργασίας πιστεύουμε ότι θα φέρει τη βιωσιμότητα και θα βοηθήσει την οικονομία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Ιζαμπέλο. Ο Σαλβαδόρ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω την άποψη της Μαρία Γράσα Καρβάλιο που είναι σκιώδη εισηγήτρια από την ομάδα μου για αυτή την έκθεση για το EIT συγκεκριμένα. Πέντε σημεία θα σας διαβάσω. Είναι η άποψή της. Ε, διότι η Μαρία Γράσα δεν μπορούσε να είναι εδώ, είναι στη ΣΥΠΑ σήμερα. Δεν μπορούσε να βρίσκεται σε επιτροπή προπολογισμό. Λοιπόν, διαβάζω στα αγγλικά. Αυτά τα πέντε σημεία τα οποία αφορούν τον ορίζοντα 2020, καταρχάς η κυρία Καρβάλιο συμφωνεί να αυξηθεί σημαντικά ο προπολογισμό ε, για την επόμενη επταετία, διότι έτσι το EIT θα προσελκύσει και κονδύλια από τον ιδιωτικό τομέα για τις δραστηριότητές του και έτσι θα ενισχυθεί η καινοτομία. Η ικανότητα της Ένωσης για καινοτομία. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις για να έχουμε κάποιες επιστροφές επενδύσεων του EIT. Θα πρέπει να βελτιωθεί βέβαια παράδοση αποτελεσμάτων με αύξηση των βιώσιμων οριδριόμενων εταιριών και διάφορες υποτροφίες. Επίσης η αριστεία πρέπει να είναι κατά τρίτον ο μοχλός για το EIT και θα προτείνει επίσης τη έβριση συμμετοχής για να διευρυνθεί η αριστεία και να εξοπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτή η αρχή των σκαλοπατιών προς την αριστεία πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή ισχυρών μονάδων στην εξαιρετική εμβριακή αριστεία. Τέταρτον, πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα απλούστευσης. Και τέλος, το EIT θα δημιουργήσει μεγαλύτερες συνέργειες και μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και μετά διαρθρωτικά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να... Α, μήπως θέλετε εσείς να πείτε κάτι κύριε Σιγητά. Ναι, γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα. Να ευχαριστήσω όλους, γιατί τα σχόλια ήταν πολύ καλά και με εκφράζουν. Νομίζω ότι όλα τα σχόλια θα τα λάβουμε υπόψη και με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας και θα μάθω πολλά, είμαι βέβαιος, από αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 17η Ιουλίου, όχι η 16η, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την υιοθέτηση της γνωμοδότησης της συνεδρίασή μας στις 6 Σεπτεμβρίου, ούτω ώστε να περάσει στην Ήτρε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και να πάει στην Ολομέλη στο τέλος του 2012. Έχουμε τρία λεφτά. η κυρία Ντεσόουζα μπορεί να πάρει το λόγο για το σημείο 20 για να μας παρουσιάσει σε τρία λεφτά το κείμενό της, όσο έχουμε τους διερμηνείς μαζί. Eh, Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξέρετε ότι η έκθεση έγινε από τον συνάδελφο Μιγγέλ Πόρτας, ο οποίος απεβίωσε τον Απρίλιο. Νομίζω ότι το ενημερωτικό δελτίο που έχουμε συνοψίζει καλά το θέμα. Εν πάση περιπτώσει θα υπογραμμίσω κάποια σημεία. Καταρχήν υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που θέλουν να καταργήσουν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και είναι παράδοξο ότι κάποια κράτη-μέλη μεταξύ αυτών εξουσιοδοτούν το Ταμείο και έχουν και πολύ ισχυρή βιομηχανία. Δεύτερον, αυτό είναι Ταμείο κατεπήγοντος, δεν είναι διαρθρωτικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει σε περίοδους κρίσης ένα τέτοιο ταμείο. Σήμερα και αύριο θα ψηφίσουμε στην ε, Ισπανία και τη Δανία γιατί υπάρχουν κατεπίγουσες καταστάσεις στις χώρες αυτές σε κάποιους τομείς. Λίγο επηρεάζει τον, τον ενωσιακό προϋπολογισμό το ταμείο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα ταμείο που μπορεί να κάνει διαφορά, τη διαφορά. Επίσης είναι σημαντικό μέσα από αυτό το ταμείο να αντιμετωπίζουμε θέματα σε συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ε, εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους, Στη Γεωργία υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν στην Επιτροπή Γεωργίας από ειδικού. Η γνωμοδότηση εδώ ε, εστιάζει την, ε, στον αποκλεισμό αυτού του τομέα της Γεωργίας ε, γιατί δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του κανονισμού. Επίσης να μιλήσω σύντομα για τον παρόντα κανονισμό που διέπει το Ταμείο η πρόσβαση στο Ταμείο είναι χαμηλή λόγω των κριτηρίων επιλεξιμότητας που κάνουν το Ταμείο λιγότερο ελκυστικό για κάποιους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος από το 2007 δεν ζήτησε βοήθεια από αυτό το Ταμείο, για παράδειγμα. Νομίζω ότι πρέπει να μειώσουμε το κατόφλι, τα οριακά τα κατώτερα όρια από 500 σε 300 άτομα εργαζόμενα σε μια επιχείρηση για να είναι επιλέξιμη να ε, υποστηριχθεί από το Ταμείο. Έτσι, κάποιες χώρες που έχουν πολλές μιμιέ θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο Ταμείο. Η υλοποίηση επίσης ήταν πολύ βραδία. 18 μήνες με 2 χρόνια είναι ο χρόνος απόκρισης καμιά φορά. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος αντίδρασης πρέπει να είναι ταχύτερος, μικρότερος. Επίσης, η επίπτωση του προϋπολογισμού. Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Προϋπολογισμού να το συζητήσει. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά ε, που, θα, ε, που έχουν δοθεί σε αυτό το ταμείο. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν 50.000 που διατέθηκαν στο Ταμείο, αλλά πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αύξηση ώστε να είναι διαθέσιμα τα κονδύλια ε, ταχύτερα και η ανταπόκριση σε αιτήματα να είναι ταχύτερη και να αποδεσμεύονται πιο γρήγορα. Πρέπει να ανταποκρινόμεθα στα αιτήματα πιο γρήγορα. Αυτές είναι οι αδυναμίες στο Ταμείο που εντοπίσαμε μαζί με άλλα μέλη της Επιτροπής. Πιστεύουμε επίσης ότι έχει πολλά καλά το Ταμείο αυτό γιατί μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε κατεπίγουσες και δύσκολες καταστάσεις και επίσης είναι ένα μέσο ευέλικτο γιατί εξατομικεύει τις λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες και νομίζω ότι οι αρετές του Ταμείου ξεπερνούν κατά πολύ τα μειονεκτήματά του και αυτό είναι κάτι που θα πω στις χώρες που θέλουν να το καταργήσουν. Τέλος, έχουμε προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 17 Ιουλίου. Δεν θα πούμε τίποτα για τις τροπολογίες ε, τώρα, προφανώς. Αλλά εγώ και η ομάδα μου θέλουμε να συζητήσουμε ε, τυχόν τροπολογίες με άλλους συναδέλφους από άλλες ομάδες και να καταλήξουμε μαζί τους από τώρα μέχρι 17 Ιουλίου, μετά τις 17 Ιουλίου ε, σε συμβιβαστικές τροπολογίες για να παραμείνει το Ταμείο αυτό ιδιαίτερα στην κρίση που ζούμε τώρα. Ευχαριστώ. Διάφοροι ζητάνε τον λόγο, αλλά ζητώ κύριε Ντάρντεν συγγνώμη από εσά γιατί είμαι υποχρεωμένο να θέσω τέρμα σε εργασία. 12.30 ώρα. Όπως είπε η κυρία Άλτα σου, Σόουζα, η ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι η 17η Ιουλίου, 12 ώρα το μεσημέρι, και την προηγούμενη έκθεση. Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση 6 Σεπτεμβρίου, υιοθετούμε την ε, υιοθέτηση στην οποία Απασχόληση τον Οκτώβριο και εν συνεχεία περνάει από την Ολομέλεια. Όλοι όσοι να πάρουν το λόγο ή να θέσουν ερωτήσεις, να το κάνουν διμερώς στο περιθώριο της συνεδριασής μας τόσο ώστε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσει σα. σας. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να παρατείνω αυτή τη συζήτηση. Σταματώ εδώ τη συνεδρίαση. Υπενθυμίζω στους συντονιστές ότι θα τα ξαναπούμε σε αυτή την αίθουσα στις 2 η ώρα. Και σε ό,τι αφορά την α, ολομέλεια της Επιτροπής Προπολογισμών, ξαναρχίζει στις 3 η ώρα για να συζητήσουμε το θέμα των οργανισμών. Το θέμα των οργανισμών. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα από τις 3 μέχρι τις 4, το θέμα των οργανισμών.